colleagues. Ah, grazie. Colleagues, can we, uh... Μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσως αγαπητοί συνάδελφοι. Can everybody please take their seats? Um, hello. Okay. Okay, colleagues, we're going to start. Πάμε αγαπητοί συνάδελφοι. Okay, colleagues, um, I've uh, been uh, συνάδελφοι να αντικαταστήσω τον πρόεδρό μας ο οποίος κολλείεται λόγω προηγουμένων υποχρεώσεων. Είμαι απροετοίμαστη πρέπει να το πω για το να προεδρεύσω σε αυτή τη συνεδρίαση. Πάντως το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ίδιας αυτής της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις, προτείνω να εγκριθεί με μια μικρή αλλαγή ή μια μεγάλη αλλαγή αν θέλετε. Α, έχετε κάποια παρατήρηση παρόλα αυτά. Κυρία Μορβάη. Νομίζω ότι σήμερα συνέβη κάτι το οποίο ήταν πραγματικά έκτακτο. Η επίθεση του Ισραήλ σε αυτούς οι οποίοι φέρνανε βοήθεια στην Γάζα είναι μια τεράστια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι και έγκλημα πολέμου Ίσως δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι συνεχίζουμε σε να μην συμβαίνει, συμβαίνει τίποτα. Νομίζω ότι εμείς ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ίσως αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στη συνεδρίασή μας. Βλέπω τους συναδέλφους, αλλά προσωπικά δεν νομίζω ότι αναπόκειται στη δική μας επιτροπή χωρίς καμία προηγούμενη προετοιμασία να δώσει μια αντίδραση. Προφανώς θα το αντιμετωπίσει η Ολομέλεια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα είναι στη μέση διάταξη ως κατεπήγον θέμα αυτό και η αρμόδια επιτροπή εξάλλου είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Χωρίς να ξέρουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τίποτα για τις λεπτομέρειες των γεγονότων και το πώς εκτιλήχθηκαν, εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εδώ κάποια δήλωση. Βλέπω πολλούς συναδέλφους να ανέβουν καταφατικά, οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Λοιπόν, η αλλαγή στη μέση διάταξη που ήθελα να προτείνω. Δυστυχώς, ο κύριος Έρικ Χόλτερ, ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ που θα συζητούσε μαζί μας αύριο το πρωί, δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει. Λυπούμαστε. αλλά φαίνεται ότι και στη χώρα του έχει να αντιμετωπίσει μερικά πολύ κατεπήγοντα θέματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο. Ω εκ τούτου, στη θέση αυτού του θέματος θα συζητήσουμε το σημείο 14 αύριο στις 10 και Αυτή είναι η γνωμοδότηση για την οδηγία σε σχέση με τα διαζύγια. Επίσης και το σημείο 15 που είναι η Συμφωνία Επανεισδοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πακιστάν που θα συζητηθεί στις 10.30. Με αυτές τις αλλαγές λοιπόν σας προτείνω να εγκρίνετε την ημερησία διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σας ευχαριστώ. Ανακοινώσει Πρόεδρου. Η γραμματεία μας εξ ονόματος του κ. Λόπες Αγιλάρ σας έστειλε μια, ένα σημείωμα την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει στον ετήσιο προπολογισμό, Ζητείτε από τα μέλη να στείλουν τι προτάσει του στη γραμματεία το αργότερο το μεσημέρι τη 5η 3η Ιουνίου. Κύριε Μπουσουτήλ, σα ευχαριστώ. Ό,τι είναι πάρα πολύ περιοριστική αυτή η προθεσμία για να μπορέσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε λογική πρόταση σε σχέση με θέματα προϋπολογισμού. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους λοιπόν να υποστηρίξουν την πρότασή μου να παραταθεί αυτή η προθεσμία τουλάχιστον για λίγες μέρες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε καλύτερα για το θέμα αυτό και όχι να χάσουμε την ευκαιρία λόγω προθεσμιών. Δεν έχω καμία προσωπική αντίρρηση, αλλά νομίζω ότι η Γραμματεία τόνισε ότι αυτή η προθεσμία οφείλεται στη διαδικασία του προπολογισμού, γιατί ε, επίκειται η συνεδρίαση τη Επιτροπή Προπολογισμών. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να παραταθεί αυτή η προθεσμία, ούτε μισή μέρα. Μήπως μπορούμε να στριμώξουμε λίγα και το χρόνο μετάφρασης για να κερδίσουμε εμείς χρόνο. Μισή μέρα κέρδισε. Μπράβο. Είδατε. Κύριε Μπούσουτιλ, πρέπει την Παρασκευή να πάει στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Μα την προηγούμενη εβδομάδα μας τα στείλατε αυτά τα email. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν μη κοινοβουλευτική εβδομάδα, πολλοί από εμάς ταξιδεύουμε εκτός Βρυξελών, όταν μας δίνετε ένα τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα, είναι σαν να μας λέτε ότι δεν μας ενδιαφέρει σαν να μου μας λέτε ότι δεν, δεν σας ενδιαφέρει τι, τι είδους προτάσεις θα κάνουμε, είτε θα μας δώσετε τη δυνατότητα και πραγματικά μια δυνατότητα ως Επιτροπή να κάνουμε κάποιες προτάσεις ή καθόλου. Αυτό είναι τώρα ανέκδοτο. Δεν μπορούμε μέσα σε δύο μέρες να έχουμε μια πρόταση για ένα πιλωτικό σχέδιο ή μια προπαρασκευαστική δράση. Όλα αυτά πρέπει να εξεταστούν σε βάθος μέσα σε κάθε πολιτική ομάδα και θα πρέπει να συζητηθούν και μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή μας, στη ΛΥΜΠΕ, ώστε να έχουμε και μία κοινή αντιμετώπιση μέσα στην Επιτροπή μας. Αλλά το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι ανέκδοτο. Συμφωνώ, αλλά το θέμα της ε, της, ε, της εβδομάδος της ε, Τυρκουάς δεν είναι επιχείρημα. Όλοι μας έχουμε κινητά τηλέφωνα και email και μπορούμε να είμαστε πληροφορημένοι. Εγώ θα πρότεινα να ζητήσουμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προεκολογισμού εάν είναι δυνατόν να έχουμε μια παράταση για την προθεσμία. Θα το ζητήσουμε σήμερα το απόγευμα για να έχουμε μια απάντηση μέχρι αύριο πρωί. Εγώ όμω θα σας ζητούσα παρόλα αυτά, εάν δεν λειτουργήσει αυτό, εάν δεν λειτουργήσει για λόγους οι οποίοι είναι διαδικαστικοί, γιατί εμείς δεν είμαστε κύριοι της διαδικασίας του προπολογισμού, αν δεν γίνει αυτό, να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη ευελιξία και να προσπαθήσουμε επί της εκτάκτου αυτής βάσης να εργαστούμε για να μην χάσουμε την ευκαιρία να καταθέσουμε τροπολογίε. Νομίζω ότι θα έχουμε ήδη κάποιε ιδέε για τα θέματα. Κάνουμε μια προσπάθεια. Κύριο Σάλβαρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλώ για να καταπραίνω τι ανησυχίε του Σίμωνο, όλε οι προτινόμενε προπαρασκευαστικέ δράσει ή τα πιλωτικά σχέδια μέσα στην έκθεσή μα θα τύχουν αντική απάντηση έτσι κι αλλιώς γιατί δεν πρόκειται με αυτή την έκθεση να πετύχουμε τίποτα. Αν θέλουμε να προωθήσουμε πιλωτικά σχέδια ή προπαρασκευαστικέ δράσει θα πρέπει να γίνει αλλού αυτό. Ο εισηγητή που έρχεται από την ομάδα του κ. Μπουσουτήλ ούτω ή άλλω διαγράφει όλε τι προτάσει για προπαρασκευαστικέ δράσει και πιλωτικά σχέδια. σω θα ήταν χρήσιμο, κ. Μπουσουτήλ, με του συναδέλφου σα να καταλάβετε καλύτερα γιατί δεν δέχεται αυτέ τι προτάσει αλλά τα πιλωτικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές δράσεις θα έρθουν σε μια μεταγενέστερη ε, έκθεση και γι' αυτό θα πρότεινε στον κύριο Μπουσουτήλ να συζητήσει πρώτα με τον εισηγητή για να δει πού ακριβώς μπορούμε να θέσουμε αυτές τις προτάσεις για πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις. Μερσή, λέει η πρόεδρος. Ίσως μπορούμε να πάρουμε μια διτή προσέγγιση για να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα ζητήσουμε και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών αν μπορεί να δοθεί λίγο περισσότερο χρόνο. Ψηφοφορίες τώρα. Φέρατε όλες τις κάρτες σας. Δεν τις φέρατε. Τότε δεν μπορείτε να ψηφίσετε, δεν μετράτε. Δεν έχουμε πολλή ώρα να ψηφίσουμε. Εκκλησία γνωμοδότηση Σταύρου Λαμπρινίδη για την διακυβέρνηση του διαδικτύου, τα επόμενα βήματα. Και υπάρχουν πολλές συμβαστικές προτάσεις, πολύ πεπλεγμένες. Υπομονή λοιπόν. Παράγραφος 1. υπάρχει ένα συμβαστικό κείμενο με αίτηση για ψηφοφορία κατά τμήματα από τους φιλελεύθερους. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρώτη παράγραφος. Διορθώνει η πρόεδρος, όχι εγκριθεί η τροπολογία, άρα πάμε στην παράγραφο 2, όχι η τροπολογία 4 έχει αποσυρθεί. Λοιπόν, τροπολογία 6 του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 7, με μια προφορική τροπολογία του εισηγητή και της κυρίας Βερζά. Συμφωνείτε όλοι να ψηφίσουμε μαζί με την προφορική τροπολογία, ωραία, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 του κυρίου Βος σε, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ο κύριος Άλβαρο. Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στη συμβαστική τροπολογία 2, μία διευκρίνηση θα ήθελα. Λέει μέσα στο κείμενο, όπως βλέπουμε στην επόμενη σελίδα, στο τέλος, ότι όταν ε, συνδυάζουμε το κυβερνοέγκλημα με την παιδοπορνογραφία. Όταν καταπολεμούμε, όχι combining, combating εννοούμε προφανώς, έτσι. Ναι, εντάξει, τυπογραφικό λάθος λέει η Πρόεδρος. Ε, συμβαστική τροπολογία 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, Α, υπάρχει νέα εκδοχή του κειμένου. Ε, θα βοηθούσε να την είχα. Μία, η νέα συμβαστική τροπολογία υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 11, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το τροποποιημένο σχέδιο γνωμόδοτης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε με μία ψήφο κατά και μία αποχή. Όχι, δύο ψήφους κατά, λέει η Πρόεδρος. Ο εισηγητής. Προφανώς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω επίσης ε, για την παράγραφο 5 τροπολογία 11 στον κατάλογο της ψηφοφορίας ότι παρότι ε, συμφωνήθηκαν σημαντικές ε, περικοπές στον προϋπολογισμό μας στην Ελλάδα ποτέ δεν δέχτηκα περικοπή στο όνομά μου. Λαμπρίνης λέει εδώ και όχι Λαμπρινίδης. Μπορείτε να το φροντίσετε. Δεν το έχει εγκρίνει αυτό η ελληνική κυβέρνηση. Η Λαμπρινίδης καμία περικοπή δεν θα περάσει. Uh, uh, Μια παρατήρηση. Καλό θα ήταν όμως, γιατί δεν χρειάζεται να τυπώνουμε τόσες πολλές σελίδε, θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Κύριε Κάσμαν, άμα, <laughs> ναι, άμα περικόψουμε το δικό σας το όνομα και γίνει Κάσ, δηλαδή μετρητά, θα είναι καλύτερα. No cash man όμως με φωνάζουν. Δεν έχω μετρητά. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο σχέδιο σύστασης για την πρόταση απόφαση του Συμβουλίου και λοιπά για τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισλανδία και την Νορβηγία για την εφαρμογή και τα λοιπά και τα λοιπά ε, του κυρίου Μπουσούτιλ. Ε, ε, δεν έχουμε τροπολογίες. Κύριε Μπουσουτήλ, ε, προσέξτε λίγο γιατί είναι το έργο σας εδώ. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, το μόφωνο. Ε, τώρα θα περάσουμε στο σχέδιο σύστασης για την πρόταση για τη συμφωνία ανάμεσα αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου του Πριγκιπάτου Λιχτενστάιν και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την συμμετοχή ε, στην επιχειρησιακή συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πω, πω. Να γιατί οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που κάνουμε. Συγητής ο κύριος Κλάς, καμία τροπολογία, μια ψηφοφορία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Κύριε Γιακουλίνο, κατά ψηφίσατε. Τι είσαστε, υπέρ ή κατά. Α, υπέρ, μάλιστα. Είμαι πολύ υπέρ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πα, τελείωσαν οι ψηφοφορίες και... Πάμε στο επόμενο σημείο εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σέγγεν όσον αφορά το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στρέφομαι στον εισηγητή μας, τον κύριο Κοέλιο. Θέλετε να κάνετε την εισαγωγική σας παρουσίαση, κύριε Κόιζα. Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έξι σημεία. Πρώτον, περί τίνος πρόκειται. Από την προσχώρησή του το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες αυτές, Ρουμανία και Βουλγαρία, Άρχισαν τις προπασκευαστικέ εργασίες για να ενταχθούν πλήρως στο χώρο Σέγγεν. Υπενθυμίζω εδώ στους συναδέλφους πως υπάρχουν διάφοροι φάκελοι που πρέπει να αναλυθούν. Προστασία δεδομένων. Το ΣΥ, Σύστημα Πληροφοριών του Σέγγεν, ε, όλα τα σύνορα, η αστυνομική συνεργασία και οι θεωρήσεις. Χρειάζεται θετική ανάλυση σε όλους αυτούς τους φακέλους. Είναι εκ των όνου Κάνεφ για να λάβει απόφαση το Συμβούλιο για να καταργήσει τα εσωτερικά σύνορα με αυτά τα κράτη-μέλη. Άρχισε η ανάλυση με αυτή την ανάλυση που συζητούμε τώρα για την προστασία των δεδομένων ε, που έγινε 27 με 30 Απριλίου του 2009 και μετά τα αποτελέσματα της ανάλυσης ε, γίνεται να αρχίσει η διαδικασία αξιολόγησης ε, για το ΣΥΣ, το Σύστημα Πληροφοριών του Σέγγεν. Αυτό συνεπάγεται μεταφορά δεδομένων από το ΣΥΣ προς αυτά τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι εκρεμεί ένα ζήτημα με το Συμβούλιο σχετικά με την διαβίβαση των εγγράφων. Τα έγγραφα θεωρούνται διαβαθμισμένα χάρη στον πρέσβη της Ρουμανίας που τον ευχαριστώ ε, καταργήθηκε η διαβάθμιση αυτών των εγγράφων και θα διαβιβαστούν σε όλους τους συναδέλφους αλλά θα έχουμε αυτό το πρόβλημα για τους επόμενους φακέλους. Επιμένω λοιπόν ώστε αμελήτη η υπογραφή ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια συμφωνία σχετική με τη διαβίβαση των εγγράφων αυτών. Το Κοινοβούλιο μπορεί να εκτιμήσει το πώς ε, το αν είναι εμπιστευτικά τα έγγραφα που έχει ήδη στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία για τα έγγραφα που στέλνει το Συμβούλιο. Τρίτον, η Βουλγαρία... Για τη Βουλγαρία εντοπίστηκαν κάποια προβλήματα για τη χρήση προσωπικών δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας. Ε, παρατηρήθηκαν ατέλειες ε, στην αρμόδια Εθνική Αρχή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Ε, και τον Ιανουάριο του 2010 κατάληξαν οι αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ακολουθήθηκαν οι σχετικές συστάσεις και τον Απρίλιο το Συμβούλιο αποφάσισε ότι υπερπηδήθηκαν όλα τα εμπόδια που είχαν εντοπιστεί νωρίτερα. Για τη Ρουμανία τώρα ε, εντοπίστηκαν ε, κάποιες ε, αδυναμίες σχετικά με δύο νόμους πάλι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως προς τους όρους λειτουργίας της Εθνικής Αρχής για την Προστασία των Δεδομένων. Το Φεβρουάριο του 2010 οι αναλυτές αποφάσισαν ότι εδώ θιέσια συνέχεια στη συστάση. Εκκρεμούν κάποια ζητήματα βέβαια, αλλά όσα ζητήματα εκκρεμούν δεν θέτουν ένα αμφιβόλο την αξιολόγηση του Συμβουλίου βάσει της οποίας είναι σε θέση η Ρουμανία να ε, ε, κάνει την ανάλυση των προσωπικών δεδομένων δυνάμει των κειμένων κανόνων προστασίας αυτών. Τέλος, Περιμένουμε την τελευταία αξιολόγηση, ε, αλλά θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να επικυρώσει τη θετική αξιολόγηση του Συμβουλίου για την ε, Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά πρέπει να απαιτήσουμε κατά τη γνώμη μου να ενημερωθεί μέσα σε έξι μήνες το Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που θα δοθεί στις ε, συστάσεις που ακόμη δεν έχουν πλήρως υλοποιηθεί. Τέλος, έκτο και τελευταίο σημείο. Ε, συζητήσαμε ήδη την αξιολόγηση του Σέγγεν και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο πέρσι τον Οκτώβρη ε, εξέδωσε αρνητική γνωμοδότηση για δύο πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη διαδικασία αξιολόγησης του Σέγγεν. Επιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέες πρωτοβουλίες. Αύριο θα συναντηθώ άτυπα με τον αρμόδιο επίτροπο για αυτό το θέμα και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω δύο σημεία που έχουν θεμελιώδη κατά μεσημασία. σημασία. Πρώτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την ιδέα δύο διαφορετικών μέτρων προτύπων ε, ανάμεσα δηλαδή στις χώρες ε, που είναι ή μέσα στο Σέγγεν ήδη και τις χώρες που είναι να προσχωρήσουν στο Σέγγεν. Οι ίδιοι οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε ολόκληρο το χώρο Σέγγεν είτε είναι υποψήφιες οι χώρες είτε ήδη έχουν προσχωρήσει στο χώρο Σέγγεν και δεύτερον υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης με παρέμβαση ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συγκεκριμένα της της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αλλά αυτό δεν αποκλεί την συμμετοχή των κρατών μελών. Όταν κάποιος μιλάει για το Σέγγεν, τι εννοεί. Δημιουργούμε ένα χώρο αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, που είναι απαραίτητη για να καταργηθούν τα εσωτερικά σύνορα και αυτό είναι ε, μια προστιθέμενη ε, αξία που πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι. Αυτά τα σχόλια ήθελα να κάνω εν είδη εισαγωγής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Κουέλιου. Πρωτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να προσκαλέσω το Συμβούλιο καθώς και την Κομισιόν να δώσουν κάποια απάντηση, κάποια αντίδραση αν θέλουν. Ο κύριος Χωσέ Μανουέλ Ροδρίγες ε, από, το Συμβούλιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η παρουσίαση της έκθεσης Κουέλιου βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ πλήρης και δίνει μια σαφή εικόνα της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Το Συμβούλιο, θέλω απλώς να σας υπενθυμίσω, έχει τον στόχο, τον κοινό στόχο, μαζί με το Κοινοβούλιο εξάλλου, να διευρύνουμε τον χώρο του Σέγγεν προς τη Βουλγαρία αλλά και τη Ρουμανία το Μάρτιο του 2011. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που Όλοι οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες αυτές, οι βουλγαρικές και ρουμανικές αρχές και η Επιτροπή ε, Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν καταβάλει προσπάθειες για να εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να γίνει η ένταξη των χωρών αυτών στο Σέγγεν ως ούπο. Είναι πολύ σημαντικό εξάλλου για το Συμβούλιο να διατηρήσει την πλήρη υποστήριξη και αρρωγή της ε, Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι θα προέλθει από εσά μια θετική γνωμοδότηση η οποία θα εγκριθεί στην επικείμενη Ολομέλεια του Ιούνιου και έτσι θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό στην διαδικασία αυτή ένταξη των χωρών αυτών στις, στο Σέγγεν, επιτυγχάνων έτσι τον στόχο που έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Επομένως, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τη συνεργασία του κυρίου Κουέλιου, ο οποίος πάντα έχει δώσει μια έντονη και συνεκτική αρρωγή στα θέματα αυτά και πιστεύω ότι και το Συμβούλιο και η Ισπανική Προεδρία πρέπει να εκφράσουν πλήρως την ευγνωμοσύνη στον κύριο Κουέλιου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μόνικα Μόσχαμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι παρούσα παρακαλώ. No, Mrs. Όχι. Κανένα άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να σχολιάσει. Ενδιαφέρον αυτό. Κανένα συνάδελφος θέλει το λόγο. Ούτε. Καλώ. α ε, επανέλθουμε στον εισηγητή, τον κύριο Κοέγια. Α, ο κύριος Έντσου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Κοέγιο, γιατί αν κατάλαβα καλά, εμείς θα εγκρίνουμε την πρόταση αυτή απόφαση. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ο εισηγητής, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στην εφαρμογή του συστήματος πληροφόρησης Schengen SIS 2 δεν είναι πρόβλημα για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για να ενταχθούν στο σύστημα καθόλου. Διότι είχαμε το σύστημα SIS 1 συν το οποίο λειτουργεί και ε, απλώς θα χρειαστεί μετάβαση στο νέο σύστημα για να αρχίσει η λειτουργία του. Και νομίζω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής μας υποστηρίζουν την έκθεση του κυρίου Κοέγιο και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, ενημερώνει, να μας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα ε, για την ένταξή μας στο Σέγγεν. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναλαμβάνουμε δράσεις και προχωρούμε σε ενέργειες που έχουν επιπτώσεις στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό που είναι καθήκον μας λοιπόν είναι ε, η προώθηση και η πρόσπιση των ευθεριών και των δικαιωμάτων τους. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι δικαίωμα που δύσκολα αποκτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά θα πρέπει να απολαμβάνουν το δικαιώματος αυτού. Και θα πρέπει να δείξουμε σύνεση και φρόνηση για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να αποκτήσουν το δικαίωμα αυτό. Δεν θα πρέπει να ορθώνουμε φραγμούς ε, στα θεσμικά όργανα μεταξύ μας, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που έχει σημασία είναι να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για ε, θέση σε ισχύ των δύο αυτών ε, κρατών. Συνένταξη του Σέγγεν δηλαδή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή, λέει εδώ ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η Δευτέρα Ιουνίου, το μεσημέρι, μεθαύριο δηλαδή. Στις 10 του μηνός θα ψηφίσει η Επιτροπή μας και η Ολομέλεια στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Ασυνήθιστα σφιχτό είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Θα μας εξηγήσετε τη σοφία σας κύριε Σιγητά γιατί προέκυψε αυτό. Madam Πράγματι κυρία Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να σεβαστούμε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το Κοινοβούλιο κατέβαλε κάθε προσπάθεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να ανταποκριθεί στην ε, ανάγκη αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία, αλλά θέλω να ζητήσω από την Προεδρία να κάνει ό,τι μπορεί για να επιληθεί το θέμα των εμπιστευτικών εγγράφων. Το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα. είχε στην αρχή προβλεφτεί ότι θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει αυτή η αποδιαβάθμιση των εγγράφων και θέλω να ευχαριστήσω επομένως τον πρεσβευτή της Ρουμανίας για το θέμα αυτό. Αλλά για τα λοιπά θέματα, για το σύστημα πληροφόρησης του Σέγγεν και τα λοιπά, άμετα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να προχωρήσουμε στην αποδιαβάθμιση εγγράφων όταν υπάρχουν στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ασθενή σημεία στα σύνορα. Είναι κατεπίγω. λοιπόν να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτά τα έγγραφα θα μπορέσουν να διαβιβαστούν στο Κοινοβούλιο γιατί είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει, δεν μπορεί να ψηφίσει σε σχέση με έγγραφα τα οποία δεν έχει στα χέρια του. Θέλω να ζητήσω λοιπόν από την Ισπανική Προεδρία να μας βοηθήσει να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό το ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι σαφές το μήνυμα αυτό και θα συζητηθεί και στη συνέχεια της μερισίας διάταξης η δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι και όλα η μοναδική περίπτωση που έχουμε έλλειψη επαρκούς διαφάνειας και διστακτικότητος από την πλευρά της Κομισιόν και του Συμβουλίου να δώσουν στη δημοσιότητα έγγραφα αυτό με φέρει στο σημείο 7 της σημερινής διάταξης, όπου πάλι και εσείς κύριε Κουέλιου, εσείς είσαστε ο, ο εισηγητής για τα συστήματα πληροφορικής στον τομέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η Κομισιό παρουσίασε τον προηγούμενο Μάρτιο μια νομοθετική πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε τον... στις 7 Απριλίου ενώπιον της Επιτροπής μας και η πρόταση αυτή θα αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας συναπόφαση όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλω να προσκαλέσω λοιπόν τον κύριο εισηγητή να κάνει την παρουσίασή του και μετά η Κομισιόν θα απαντήσει και θα υπάρξει συζήτηση. Κύριε Κουέλιου. Ευχαριστώ. Ε, συναντήθηκαμε με, με τους σκιώδεις εισηγητές για να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκπονούμε τις εκθέσεις ώστε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εγώ ζήτησα γνωμοδοτήσεις χωρίς έκθεση. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα. Φαίνεται να είναι αυτή η επιθυμία των μελών της Επιτροπής μας. για να ε, καταλήξουμε στην ευρύτερη δυνατή συνένεση ε, στην Επιτροπή μας. Πρώτο σημείο. Πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, αποφάσισε η Επιτροπή τελικά να υποβάλει μία μόνο πρωτοβουλία. Εμείς ζητήσαμε από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αν αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος για να εξετάσουμε αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Γιατί, διότι δημιουργείται πρόβλημα ως προς τη συμμετοχή κάποιων κρατών μελών. Δεν εμπλέκονται στον ίδιο βαθμό όλα τα κράτη-μέλη στα διάφορα εργαλεία, ΣΥΣ, ΒΙΣ, Eurodac. Άρα είναι μάλλον προφανές ότι δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα για συμμετοχή στα ε, επιμέρους συστήματα. Ακόμη δεν έχω λάβει τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και αυτό είναι ένα από τα εκρεμή προβλήματα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Δεύτερον, η υπηρεσία Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι επικρίνουν την ιδέα σύστασης νέου, νέου οργανισμού. Μα θα σας θυμίσω ότι το ίδιο το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει ε, υπηρεσία που θα ειδικεύεται ε, για την επιτέλεση αυτών των καθηκόντων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα που ζήτησε ε, ε, τη σύσταση του οργανισμού το Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη και η μελέτη αντικτύπου κατέδειξε ότι από πλευράς προϋπολογισμού είναι επίσης η καλύτερη δυνατή λύση. Υπήρχαν και άλλες εναλλακτικέ λύσεις, θα θυμάστε. Κάποιες είχε ήδη απορρίψει το Κοινοβούλιο Παραδείγματο χάρη, η ιδέα να ε, παρέμβουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη διακυβερνητική διαχείριση όπω σήμερα ή να χρησιμοποιήσουμε τη Europol, το Frontex ή κάποιον άλλο υπάρχοντα οργανισμό και να χρησιμοποιήσουμε το δικό του δυναμικό για τη διαχείριση των συστημάτων. Αυτό δεν αποδε... μπορεί να είναι αποδέκτο από πλευράς προστασίας των δεδομένων. Δεν μπορεί ε, ένας οργανισμός να παρέχει και να καταναλώνει, να χρησιμοποιεί και να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα λόγω των κανόνων προστασίας αυτών. Οπότε η σύσταση νέου οργανισμού είναι η βέλτιστη δυνατή λύση, κατά τη γνώμη μας. Πλην όμως ε, πρέπει να ρυθμίσουμε διάφορα προβλήματα. Πρώτον, ο οργανισμός ε, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται νέα συστήματα όπως το Ευρωπαϊκό PNR ε, ή το Ευρωπαϊκό Σύστημα για τις Καταχωρήσεις. Για να διαχειριστεί νέα συστήματα αυτός ο οργανισμός πρέπει να έχουμε ένα νέο νομικό μέσο που υπάγεται στη διαδικασία της συναπόφασης. Τι σημαίνει αυτό. Κανένα άλλο θεσμικό όργανο, ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να διευρύνει το πεδίο του οργανισμού χωρίς να ψηφίσει πρώτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δώσει τη συγκατάθεσή του. Επίσης, ε, χρησιμοποιούνται όροι όπως ε, ε, μεγάλα συστήματα πληροφορικής, μεγάλης κλίμακας, ε, μάλλον η επιχειρησιακή λειτουργία και πρέπει να διευκρινίσουμε όλη αυτή τη φρασιολογία που χρησιμοποιείται μέσα στο νομοθέτημα για να είμαστε σαφέστεροι. Επίσης, οι στόχοι και τα καθήκοντα του οργανισμού πρέπει να προσδιοριστούν έτσι περαιτέρω. Για τα ε, πιλωτικά προγράμματα, η απόφαση ε, μέσα από αυτά τα προγράμματα, ε, να, ε, μάλλον η απόφαση για να χρησιμοποιηθούν τέτοια προγράμματα ε, δεν πρέπει να σημαίνει ότι δεν θα έχει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων του Κοινοβούλιο για τη χρήση αυτών των συστημάτων. Επίσης πρέπει να έχουμε αξιωματούχο προστασία των δεδομένων, έναν άλλον που θα είναι αρμόδιος για την ασφάλεια και τέλος έναν αξιωματούχο για τα λογιστικά θέματα. Επίσης πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να, να φροντίσουμε τα δικαιώματα ψήφου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο Είναι απαράδεκτο ένα κράτος μέλος ε, που δεν συμμετέχει πλήρως σε όλα αυτά τα προγράμματα να ε, μπορεί να ε, εκλεγεί στη θέση του Προέδρου του εκτελεστικού διευθυντή αυτού του οργανισμού. Και το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα ψήφου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρωθεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων. Οφείλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου να κατοχυρώσουμε την διαφάνεια και να μεριμνήσουμε ώστε να εφαρμοστούν πλήρω οι κανόνε προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέλο, Πρόεδρε, υπάρχει και ένα πρόβλημα ε, για την, ε, την έδρα του ε, οργανισμού. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Οπότε, εάν το Συμβούλιο συμφωνήσει για μία ε, ε, λύση αποδεκτή από το Κοινοβούλιο, εμείς δεν πρόκειται να ε, δημιουργήσουμε προβλήματα σχετικά με την επιλογή του Συμβουλίου. Είναι θέμα συναπόφασης κατά τη γνώμη μας. Ε, πρέπει να προβλέπετε μέσα στη νομική πράξη ε, και είμαστε, θα προτιθέμεθα να υπερψηφίσουμε την απόφαση του Συμβουλίου αρκεί να τηρούνται και οι αρχές που θα θέσουμε. Τι εννοώ. Θα θέσουμε διάφορες αρχές που πρέπει να τηρηθούν κατά τη γνώμη μας, παραδείγματος χάρη αν η απόφαση για την έδρα θέτει σε κίνδυνο την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια, την προστασία, αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Αν όμως στηριθούν όλες οι αρχές, τότε, κατά τη γνώμη μας, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δεχτεί την απόφαση που θα έχει λάβει το Συμβούλιο σχετικά με την έδρα ε, του οργανισμού. Λοιπόν, Για να κλείσω την παρουσίασή μου, ζητώ από τους συναδέλφους ε, να ε, συνεισφέρουν με τις απόψεις τους, ε, αν έχουν εντοπίσει άλλα στοιχεία μέσα στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λείπουν από την γνωμοδότησή μου και να με επικουρήσουν στη σύνταξη του σχεδίου έκθεσης, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να μπορέσουν να υποβάλουν στους συναδέλφους το σχέδιο. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο, αν είναι κάποιος παρόν, ε, και μετά ε, στους συναδέλφους. Ε. Η κυρία Κλάιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν απατώμε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον εισηγητή. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η προσέγγιση του. Επίσης ε, έγιναν ανταλλαγέ απόψεων και σε διάφορε επιτροπές. Είναι πολύ ε, διαφωτιστικά αυτά και επικοδομητικά για τη θέση του Κοινοβουλίου. Είδαμε και τις ε, τροπολογίες ε, του κυρίου Μαρινέσκου στην Επιτροπή Ελέγχου ε, του Προϋπολογισμού, επίσης πολύ επικοδομητικές και μπορούμε να τις δεχτούμε διότι η πλειονότητα των τροπολογιών αυτών ενισχύει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εμπλουτίζει μάλιστα. Τώρα, για τις λεπτομέρειες στις οποίες αναφέρθηκε μόλις ο κύριος Σκοέγιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει αυτή τη στιγμή ότι Πολλές από τις ανησυχίες ε, του ε, εισηγητού έχουν ξεπεραστεί, έχουν λυθεί μετά από συνεννόηση με το Συμβούλιο και πάντα σε επικοδομητικό πνεύμα και περιμένουμε την έκθεση του εισηγητού για, για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Το σχέδιο της έκθεσης. Η Πρόεδρος, θέλει να μιλήσει κανείς από το Συμβούλιο. Είναι παρόν το Συμβούλιο καταρχήν. Όχι, ορίστε. Συγγνώμη, δεν σας γνωρίζω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου θα ήθελα να σας δώσω ορισμένα στοιχεία μου επιτρέπετε για το πώς έχει η πορεία των ε, συζητήσεων και των διαβουλεύσεων στην ομάδα εργασίας. Η τελευταία συνεδρίαση της Ισπανικής Προεδρίας ε, διεξήχθη σήμερα το πρωί για τα ζητήματα του Σέγγερν, γιατί αυτή είναι η αρμόδια επιτροπή. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι με αναμονή της έκθεσης του εισηγητού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή των εισηγητών, η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου κατάφερε σε ορισμένα από τα δύσκολα και περίπλοκα κείμενα μια συμφωνία επί της αρχής ε, που συμφωνεί πολύ με τα όσα πολύ σωστά ε, επισήμενε ο κύριος ε, Κοέγιο. Αυτό που θέλουμε είναι, ένα αποτελεσματική ε, και σκόπιμη η υπηρεσία αυτή και από τη Διοργανική Συμφωνία του 2006 και η υπηρεσία, καλύτερα ο οργανισμός, θα έρθει να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη και να λύσει ε, αυτό το πρόβλημα διαχείρισης των μεγάλων συστημάτων προφορικής. Δεν υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και το Συμβούλιο αυτό που θέλει είναι να συμφωνήσει ακόμα κατά τη διάρκεια ε, της πρώτης ανάγνωσης. Τώρα όσο για την έδρα, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι προς στιγμή δύο είναι υποψηφιότητες. Μία είναι γαλλική για το Στρασβούργο και η Εσθονία προτείνει το Ταλίν. Είναι και μεγάλα τα τεχνικά ζητήματα. Το Συμβούλιο ακόμα δεν έχει υπόψη του να ασχοληθεί με το θέμα της έδρας μέχρι να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα νομικά κύματα και για το διατακτικό ή να προχωρήσει αν τι άλλο. Από την αρχή η Προεδρία ήταν σε επαφή με τον εισηγητή και τις επόμενες ημέρες ε, θα ξανασυζητήσουμε μαζί του. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να διευκολύνουμε την κατάσταση και όχι ε, να φέρουμε νέα εμπόδια. Ο εισηγητής είπε ε, το ζήτημα ε, το, της των ψήφων είναι μια μεταβλητή γεωμετρία και προς το πάνω αυτό μπορώ να σας πω μόνο και έχει να κάνει με ορισμένα κράτη-μέλη στην Ένωση. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει τρία μέλη τον λόγο. Δεν ξέρω κάποιος άλλος θέλει να προσθεθεί στον κατάλογο, τον κλείνω. Oui, merci, Madame la Présidente. Euh, je voulais... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέγιο που μπόρεσε μέσα από τις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών να καλύψει το θέμα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις προτεραιότητες της πολιτικής μου ομάδας, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Να επαναλάβω την θετική μας γνώμη για τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να είναι μια λειτουργική υπηρεσία και τα συγκεκριμένα συστήματα δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από ιδιωτικές εταιρείες με ό,τι αυτό σημαίνει σε επίπεδο ασφαλείας. Ένα δεύτερο θέμα, σύντομα πάντα, γιατί σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Κοΐο, είναι το θέμα της ενσωμάτωσης σε αυτή τη λειτουργική υπηρεσία ενός συντονιστή προστασίας δεδομένων. Ένα τρίτο σημείο, μια τρίτη προτεραιότητα είναι το εύρος αρμοδιοτήτων και ευθυνών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κάθε μορφή και δυνατότητα κατάχρησης και να περιοριστούμε σε λειτουργίες αποκλειστικά τεχνικής φύσεως. Μια τελευταία προτεραιότητα που συζητήθηκε και από τον ίδιο τον κύριο Κοέγιο και από τους ε, ισχυώδεις εισηγητές, κάθε πιθανή διεύρυνση της ε, αρμοδιότητας των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας αυτής δεν μπορεί να περάσει παρά μόνο μέσω εγκρίσεως κοινοβουλευτικής και εννοώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τελευταίο θέμα. Ε, Προφανώ δεν μπορώ να το αποφύγω, Γαλλίδα είμαι, το περιμένετε. Πράγματι θα πρέπει να προωθήσουμε μια συγκεκριμένη επιλογή, μια συγκεκριμένη πόλη, κάτι το οποίο είναι αρκετά σύνθετο βέβαια. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε ε, σε σχέση με τις δυνατότητες διασφάλισης της ασφάλειας της λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οπότε εδώ το σχετικά αποκεντρωμένο ίσως σαν στοιχείο να μην είναι το ε, θετικότερο. Εν πάση περιπτώσει είμαστε στη διάθεσή σας και θα πάρουμε μέρος στην τελική διατύπωση της εκθέσεώς σας. Ο κύριος Αλβάρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω τη χαρά να παρακολουθώ την έκθεση αυτή για την ομάδα μου και από την Επιτροπή εσωτερικών και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Και ε, έχω συνηθίσει να συνεργάζομαι με τον κύριο Κοέγιο. Είναι πραγματική χαρά αυτή η συνεργασία. Ε, αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα διευκρινίσουμε γιατί ο χρόνος είναι σύντομος. Μόνο έμεσα μπορούμε να ε, μιλήσουμε για τα θέματα είναι το ΒΙΣ και το Eurodac, τα γνωρίζετε αυτά, και το SIS2, ε, που είναι η μετεξέλιξη του συστήματος ε, πληροφόρησης στο Schengen. Τώρα, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε να έχει περάσει το σύστημα στο SIS2 και να έχει στηθεί και μετά να δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός ή όχι ή παράλληλα να στήσουμε αυτό τον οργανισμό που να διαχειρίζεται το σύστημα ήδη από το πρώτο και κάποια στιγμή θα γίνει μετάβαση στο δεύτερο. Αυτό δεν ξέρω, είναι συζητήσιμο. Ούτε ε, ποια είναι η χρονική σειρά. Ελέγχεται και αυτό. Τώρα, κάτι άλλο που ακούσαμε. Ποιος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις τράπεζες δεδομένων και των στοιχείων που ήδη υπάρχουν στο Eurodac. Ας πούμε, η Ευρωπόλ θα έχει πρόσβαση στο Eurodac. Μέχρι τώρα αυτό δεν υπήρχε, δεν ε, προβλεπόταν και θα πρέπει να το προσέξουμε. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κεντρική διαχείριση. Βεβαίως, όχι κεντρική διασύνδεση, έτσι, προσοχή. Cross references το λένε αυτό, να είναι ε, μια δέσμη ε, ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το αρχείο και ποιος θα το διαχειρίζεται. Και τώρα ε, το είπε και ο Κοέγιος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ε, ότι εκεί μπορούν να ενταχθούν και άλλες βάσεις δεδομένων στη ε, δικαιοσύνη και στο τομέα των εσωτερικών. Τι θα πει αυτό, γιατί το λένε έτσι πολύ ξερά και πολύ στεγνά και δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Ε, να, το παρακολουθούμε κι εμείς αυτό το θέμα στην Επιτροπή μας, αν θέλουν να διευρύνουν την Τράπεζα Δεδομένων. Κάτι άλλο που θα μπορούσε ίσως να απαντήσει το Συμβούλιο ή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το έχουν συζητήσει. Αυτό είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα κέντρα έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από πλευρά δεδομένων και από πλευρά πληροφοριών που θα συλλέγονται εκεί. Για την ασφάλεια με ενδιαφέρει τώρα το δεδομένο. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ε, μία ε, υπηρεσία, ένας οργανισμός να υποπτεύει κάποιον άλλον. Αλλά όταν θα μιλήσουμε για την ΕΝΗΣΑ και τη νέα εντολή που όλο και περισσότερο διαχειρίζεται και αξιολογεί ε, αυτά τα συστήματα και μπορεί να γίνει και επιχειρησιακή, ε, κάπου να εποπτεύει και αυτή εδώ την ε, υπηρεσία των οργανισμών πληροφορικής. Γιατί διαφορετικά, γιατί δημιουργούμε τέτοιες υπηρεσίες τύπου ενίσα από τον προπολογισμό προτείνουμε να μπει στο αποθεματικό, γιατί είναι 120 εκατομμύρια για μία τριετία, με βάση ε, τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εκεί έρχεται να προσθεθεί και ένας επόπτης δεδομένων, ένας εσωτερικός ελεγκτής, αυτό μπορεί να μεταβάλει το κόστος. Γι' αυτό θεωρούμε σκόπιμο στην Επιτροπή Προπολογισμών τα χρήματα να μπουν στο αποθεματικό και να χρειάζεται αιτιολόγηση για να αντιληθούν. Για να δούμε πώς θα στηθεί και η δομή αυτού του οργανισμού και πώς θα έχουν οι δαπάνες της. Αυτό το διαπιστώνει κανείς μόνο στο τέλος της έκθεσης, αν ξέρεις και το οργανόγραμμα και την αποστολή τους. Για την έδρα συμφωνώ με τον Κοέγιο. Αυτό είναι βασικά θέμα του Συμβουλίου να το συζητήσει. Αν το βάλετε στο Στασβούργο υπάρχει και κτίριο ελεύθερο. Δηλαδή ε, έχουμε χώρο. Μια φορά το μήνα πάμε εκεί, αλλά αν θέλετε για τις υπόλοιπες εβδομάδες έχουμε εγκαταστάσεις. Αλλά και η Εσθονία έχει πολύ μεγάλη πείρα με την ε, ασφάλεια των ε, συστημάτων προφορικής ε, και ε, συστήματα του ΝΑΤΟ ασφαλείας δεδομένων μετά και από την διαδικτυακή επίθεση που δέχτηκε η Εστονία στον κυβερνοχώρο, θυμάστε παλαιότερα, τα έχουν κλειδώσει αυτά. Ευχαριστώ η κυρία Ένστ και ο κύριος Άλμπρεχτ τελευταίος, εκτός αν θέλει κι άλλο το λόγο. Όχι. Η κυρία Ένστ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι έχω ησυχάσει λίγο και με ανακούφισε αυτό που άκουσα από τον κύριο Κοαΐα. Είναι πολύ στριφνό το πρόβλημα. Ε, συμφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί σας, <laughs> πράγμα που με εκπλήσει και μένα την ίδια, αλλά με χαροποιεί κιόλας γιατί ε, θα ήθελα να σας πω ότι κατά βάση συμφωνώ να σας αναφέρω όμως μερικά προβλήματα που με απασχολούν και με ανησυχούν. Ε, πρώτον, δεν συμφωνούν πολύ με αυτό. Έγιναν ε, συζητήσεις για διάφορες εναλλακτικέ προτάσεις για το πώς θα διαχειρίζεται και ποιος θα διαχειρίζεται αυτό το σύστημα. Και σχετικά ε, προφανές ε, και αυτονόητο φάνηκε να δημιουργηθεί ο οργανισμός. Εγώ θα σας έκανα και άλλες προτάσεις. Γιατί έχουμε μια πρωτοφανή τώρα συγκέντρωση, ένα συμπίλημα εκατομμυρίων ε, στοιχείων και δεδομένων. Μπορεί να ακούγεται αυτό αποτελεσματικό, αλλά να έχει και κινδύνους. Και για μας πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται η σωστή ανταλλαγή πληροφοριών, όχι αδιάκριτη ανταλλαγή και ο καθένας να έχει πρόσβαση και να τα διαχειρίζεται όπως θέλει. Και δεν με ενδιαφέρει, δεν, μάλλον δεν μου χρησιμεύει πάρα πολύ να μου λέτε ότι ο επόπτης ε, προστασίας ε, δεδομένων ε, τα ελέγχει αυτά ή έχει δικαίωμα ελέγχου. Και όταν ε, αποφασίζουμε διάφορες απαγορεύσεις, αυτές πάλι μπορούν να αναιρεθούν. Ο οργανισμός είναι ξεχωριστό ε, υποκείμενο ε, δικαίου, ξεχωριστή οντότητα, ε, αλλά τι γίνεται με τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επαναπαυθεί σε μια έκθεση πεπραγμένων ή μήπως θα πρέπει να καλούμε και τον εκτελεστικό διευθυντή να τον ακούμε. Γιατί δεν ξέρω, κάπως πρέπει να παίζει μεγαλύτερο ρόλο το Κοινοβούλιο. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι η αποστολή του οργανισμού. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τα καθήκοντά του. Ε, διαχωρισμός του συστηματος ε, ε, cs SES2, VIS και Eurodac, εντάξει, και να μην τα ανακατέψουμε όλα τα δεδομένα στο ίδιο τσουβάλι. Θυμάστε τη συζήτηση που κάναμε για το SIS2, έτσι. Είναι πολύ διχασμένη η Επιτροπή μας για αυτό το θέμα. Δεν συμφωνούμε. Στη δική μου χώρα το ΣΥΣ 2 περίπου το έχουν εξεγράψει και σκέφτονται άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Και εμείς θεωρούμε αυτονόητο ότι το ΣΥΣ 2 θα φτάσει κάποια στιγμή. Νομίζω αυτό είναι πολύ θαραλέο, για να μην το πω διαφορετικά. Δεν είναι απόλυτο, ξέρετε, ότι θα περάσουμε στο σύστημα αυτό. Άλλο θέμα. Δεν θα πρέπει να είναι λευκό επιταγή για άλλα συστήματα πληροφορικής, να πολλαπλασιάζονται τα συστήματα αυτά ε, έτσι ανώδυνα χωρίς να το έχουμε συζητήσει εμείς. Όχι. Δηλαδή να μην τους δώσουμε το ελεύθερο και να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε μια διατύπωση να περνάει μέσα από την Επιτροπή μας αυτό. Γιατί έτσι όπως το λέει δεν με ικανοποιεί. Έδρα. Ε, πάλι μη γελιόμαστε. Εκεί να δείτε καυγάς που θα πέσει και ούτε έχει λήξει αυτό γιατί υπάρχουν τεράστια διαφορετικά συμφέροντα, ούτε ξέρω αν είναι σκόπιμο να είναι μία η έδρα και να τα έχουμε συγκεντρώσει όλα σε ένα σημείο. Εντάξει, πολύ αισιόδοξα τα λέτε, αλλά τα προβλήματα παραμένουν μεγάλα και ε, ανεπιλήτα. Ο εκτελεστικός διευθυντής επίσης διαπιστώνω ότι είναι ο κυρίαρχος, έτσι, μάστερ. Και πώς θα ορίζεται αυτός. Αν συμβαίνει, αν είναι τόσο μεγάλη η εξουσία του, δεν μπορεί να διορίζεται με τον τρόπο που προτείνεται. Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό σε βάθος, γιατί είναι πολύ μεγάλη θέση και πολύ κρίσιμη. Τα ένδικα μέσα. Τι γίνεται εδώ. Αν κάποιο, α πούμε, φύγεται, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, το ψάξα, δεν βρήκα τίποτα. Και για το κόστος, ε, ε, ακούστηκε αυτό το επιχείρημα, να πω και κάτι για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα. Αν δημιουργήσουμε τέτοιο σύστημα, με τέτοια μάζα, με τέτοιο όγκο και συγκέντρωση πληροφοριών, τότε πιστεύω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διευρυνθεί στενάρα, αίσθητα, δεν ξέρω πώς και αυτό το συζητούμε, δεν αρκούν κάποιες εκθέσεις που θα κάνουμε αιτήσει, ξέρω εγώ, όχι. Χρειάζεται ουσιαστικός έλεγχο του Κοινοβουλίου και βελτίωση. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Albrecht. Ευχαριστώ. Σύντομα σχετικά γιατί επανειλημμένα έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Οι παρατηρήσεις μέχρι τώρα είναι για μένα πολύ χρήσιμες και πολύ σημαντικές. Ε, επιτρέψτε μου να επιμείνω σε κάτι που όντως ακούστηκε ήδη, αλλά θέλω να το ξαναπώ κι εγώ, ε, που είναι η διασύνδεση η διασταύρωση των ε, τραπεζών ε, δεδομένων και η χρήση από τους διάφορους ενδιαφερόμενους. Θα πρέπει αυτό να είναι ορισμένο από την αρχή και όχι εκ των υστέρων να το ορίσει ο οργανισμός. Όχι, το κοινοβούλιο από την αρχή να ξεκαθαρίσει ποιος θα έχει πρόσβαση που. Γιατί όταν συλλέγεις κάποια στοιχεία θα πρέπει να τα συλλέγεις στοχευμένα για μια συγκεκριμένη χρήση και όχι τα έχω μαζέψει και θα δω τι θα τα κάνω. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Και όσο μεγαλύτερε είναι οι βάσει δεδομένων και όσο μεγαλύτερο είναι ο όγκος των πληροφοριών που μπορούν να διασυνδεθούν, να, να συνδυαστούν, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος καταχρήσεων ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από το σκοπό που είχαν συλλεγεί. Και θα πρέπει να το πούμε αυτό όταν γνωμοδοτούμε για τον οργανισμό αυτό πληροφορικής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, μόνο με σαφή διαχωρισμό το στοιχείο και όλα τα υπόλοιπα να τα ξανασυζητάει και να τα αποφασίζει το Κοινοβούλιο. Uh, Ευχαριστώ για τη συντομία σα Ο εισηγητής θα ήθελε να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και την υποστήριξή τους. Θα ολοκληρώσω τη σύνταξη της έκθεσης στο τέλος της εβδομάδας. Θα έχετε το πρώτο κείμενο πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε να εργαστούμε από κοινού σύντομα. Να συμπληρώσω σε αυτά τα οποία ακούστηκαν το εξής εμείς θα δημιουργήσουμε μία υπηρεσία η οποία θα διαχειρίζεται τις τράπεζες δεδομένων, τις βάσεις δεδομένων. Όχι να αποφασίζει για τον τρόπο με τον οποίο τα συγκεκριμένα δεδομένα θα καθίστανται προσβάσιμα από τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο κάθε συγκεκριμένης τράπεζας δεδομένων. Αν θέλουμε σαν παράδειγμα να ανοίξουμε το Eurolat, το VIS σε άλλες υπηρεσίες, αυτό δεν θα γίνει μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά μέσω της αλλαγής του νομικού πλαισίου με το οποίο λειτουργούν οι προηγούμενες υπηρεσίες. Η υπηρεσία λοιπόν την οποία θα δημιουργήσουμε δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα, απλά δημιουργεί ένα δίκτυο δεδομένων, ένα δίκτυο μάλλον ασφαλείας, διασφαλίζει την αξιοπιστία του δικτύου μεταφοράς και ε, ενημέρωσης των δεδομένων αυτών, αλλά δεν θα έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα. Αυτό είναι προς το συμφέρον ακριβώς της προστασίας του χαρακτήρα των συγκεκριμένων δεδομένων. και πρέπει να διαχωρίσουμε πλήρως τις αρμοδιότητες τις οποίες θα έχει η συγκεκριμένη υπηρεσία με τα νομικά χαρακτηριστικά των βάσεων δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο κόρπους αυτό. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα κυκλοφορήσει το πρώτο σχέδιο, το πρόχειρο της έκθεσής μου και νομίζω ότι θα υποφεληθώ για μια ακόμη φορά από τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ κύριε Κοέγιο. Περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Θα ακούσουμε ότι μας πει ο εισηγητής μας, ο κύριος Κάσμαν. Πρόκειται για μια κοινή έκθεση της ΛΥΜΠΕ και της ΑΦΚΟ. Ο δικός μας εισηγητής είναι ο κύριος Κάσμαν. Η κυρία Γιατεμάκη είναι η εισηγήτρια στην ΑΦΚΟ. Η παρουσίαση που θα γίνει σήμερα βασίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 για την αναδιατύπωση ε, του 1049, του κανονισμού 1049 σχετικά με την πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι θα πρέπει να εμείνει στην πρόταση του 2008 ως έχει παρά τις νέες νομικές αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει εν τω μεταξύ μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, όλες οι υπηρεσίες, οι εξωτερικές και εσωτερικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιδιώκουν και την εμπιστευτικότητα αλλά και τη διαφάνεια όπως ορίζεται από τον κανονισμό 1049. Θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων αύριο με κάποιες από τις υπηρεσίες και τα όργανα τα οποία μετέχουν στην πρόταση αυτή έτσι ώστε να καταστήσουμε τα όργανα αυτά ικανά να εκφράσουν και τις δικές τους απόψεις. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχετε απολύτως δίκιο όταν λέτε πως ε, θα γίνει ακρόαση με τους εκπροσώπους των διαφόρων οργανισμών αύριο το απόγευμα και δηλώνω ικανοποιημένος διότι για να πραγματοποιηθεί αυτό εργάστηκε σκληρά, πολύ σκληρά η γραμματεία. Επίσης θα υπάρχουν και μέλη της Επιτροπής Ταγματικών Υποθέσεων στην ακρόαση. Μας απασχολεί εδώ και καιρό το ζήτημα και από την αρχή της νέας θητείας Έκανα διάφορες ε, συνεδριάσεις, ε, συναντήσεις με τους ε, συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές και το σχέδιο ε, που υπέβαλα είναι προς συζήτηση. Ο σκοπός να τροφοδοτήσει τη συζήτηση. Ε, είναι ε, προφανής οι περισσότερες τροπολογίες. Να διευκρινίσω, όταν μιλάμε για την κατάργηση του άρθρου 9 που έχει σχέση με την πρόσβαση στα ευαίσθητα έγγραφα, όπως ονομάζονται, ε, αυτή ήταν μια ιδέα που προέκυψε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο από το 1999 έως το 2001 και πρόκειται για, ε, τις, ε, για τα διαβαθμισμένα έγγραφα. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες, τώρα υπάρχουν τέσσερις πλέον, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, σχετικά με το άρθρο 9 και το θέμα των διαβαθμισμένων εγγράφων, ε, περί πρόκειται. Για να υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα όλων των θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών και των οργανισμών πρέπει να υπάρχει συνοχή. Μπορεί να μην προβλεφθούν όλες οι διατάξεις ε, της ε, πρόσβασης μέσα σε αυτό τον κανονισμό Ήδη γίνονται εργασίες για ένα μοντέλο στο Συμβούλιο που μου φαίνεται καλό. Οπότε καλό θα ήταν να έχουμε το ίδιο σύστημα ταξινόμησης σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις επιμέρους υπηρεσίες και οργανισμούς. Είπατε, Πρόεδρε, στην ε, εισαγωγή σας παρουσίαση ότι η προσέγγιση μας, και μην ξεχνάτε ότι είχε γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, η προσέγγιση μας ε, λοιπόν ευθυγραμμίζεται με την Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέκυψε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Λάβαμε υπόψη επίση την νομολογία, τη μεταγενέστερη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο νέο κανονισμό πρέπει να υπάρχει ένα συνεχτικό, ολικό, σφαιρικό, νομικό πλαίσιο που θα διέπει όλα τα έγγραφα που πρέπει να τύχουν διαβάθμιση προ συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά, όταν διαβαθμίζεται ένα έγγραφο, αυτό σχετίζεται επίση και με τον ε, περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάση του άρθρου 52 τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Άρα, ε, θα πρέπει να ε, διευκρινίσουμε αυτό το σημείο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει στις συζητήσεις που θα έχουμε με τους συνομιλητές μας. Ε, η κυρία Γιατεμάκη θα έρθει φυσικά αύριο. Θα, θα εκπροσωπηθεί και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Ε, επίσης, ο κύριος Χούστινγκς, ο επόπτης των προσωπικών δεδομένων, θα παρέμβει και ο συντονιστής για την τρομοκρατία καθώς και ένας εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και ε, θα ε, εκπροσωπείται και ε, θα έρθει ο κύριος Πίτερσα που είναι ο αρμόδιος από το Εθνικό Γραφείο της Γερμανίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και διάφοροι άλλοι. Έχω υψηλές προσδοκίες για την αυριανή συνάντηση. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία τους. Δεν επικρατεί πάντοτε ομοθυμία γιατί υπάρχουν διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις σχετικά με ε, το θέμα της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα. Το πρόβλημα είναι ότι στο Συμβούλιο δεν υπάρχει και πολύ όρεξη να εγκριθούν αυτές οι προτάσεις που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας και δεν νομίζω να αλλάξει η κατάσταση. Βέβαια, αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι να δω η νέα κυβέρνηση συντηρητικών φιλελευθέρων του Ηνωμένου Βασιλείου πώς θα τοποθετηθεί στο Συμβούλιο για να ε, μιλήσω και για την αγγλική πραγματικότητα. Ο νέος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κάμερον, είπε ε, προσωπώντας φυσικά τον, ε, τον συνασπισμό φιλελευθέρων συντηρητικών, ότι θα ε, υποστηρίξει την μεγαλύτερη ελευθερία, μεγαλύτερη διαφάνεια, με καλύτερη πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, οπότε πραγματικά ανυπομονώ να δω πώς θα τοποθετηθεί στο Συμβούλιο. Ο συνάδελφος μου, κυρίως Μέιζα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσης βλέπω είναι εδώ, έχουμε συνεργαστεί επί σειρά ετών και Νομίζω ότι στην Επιτροπή ε, θεωρούν ότι υπερβαίνουμε την εντολή μας, ε, ότι θα έπρεπε να ασχοληθούμε μόνο με το αναθεωρημένο σχέδιο και ο προηγούμενος πρόεδρος της Επιτροπή ΛΥΜΠΕ κοινοποίησε επίσημα στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να ε, περιοριστούμε ε, βάσει της διαθεσμική συμφωνίας στο αναθεωρημένο σχέδιο, διότι δεν τηρήθηκαν οι αρχές που είχαμε θέσει και άρα ο προηγούμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας έδωσε την έγκριση να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες μας Ε, και στην ε, τελική πρώτη ανάγνωση τελικά όμως δεν έγινε ψηφοφορία. Η αρχή ε, πάντως δεν ακολουθήθηκε να ασχοληθούμε μόνο με το αναθεωρημένο σχέδιο. Ε, τέλος, ε, νομίζω πρέπει να τονίσω υπόψη των συναδέλφων ότι είναι ευαίσθητες και οι τροπολογίες. Ε, οι σκιώδεις εισηγητές ε, μου ξεκαθάρισαν ότι όταν μιλώ για information πληροφορίες και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και τις πληροφορίες που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων μπορεί ε, ε, εξωτερικοί εμπλεκόμενοι φορείς να το εκμεταλλευτούν, ούτω ώστε να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που σχετίζονται με τις υποθέσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, οι προσωπικές ε, φυσικά υποθέσεις καλύπτονται από την Οδηγία Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Αλλά όταν ε, μιλάμε για προσωπικό έξοδα κτλ. κτλ οφείλω να πω στους συναδέλφους ότι όντως αυτός ο όρος information μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να τον εκμεταλλευτούν μέσα στον κανονισμό δεν θέλω κανείς στο πέρα της διαδικασίας να έρθει να μου πει δεν είχα επίγνωση αυτού του κινδύνου. Ε, δηλαδή ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος ε, να ε, υπάρξουν να, θελημένα και μη να γίνει κατάχρηση αυτού του όρου. Στις σχέσεις μας με τους εκπροσώπους των κρατών μελών, μιλάμε για κοινοβουλευτικά σώματα, μη κυβερνητικού οργανισμούς, ε, δημοσιογράφους, ε, πρέπει να, ε, προσέξουμε να μην υπάρξει συκοφάντηση ή παραπληροφόρηση που θα βλάψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία που ήθελα να σχολιάσω. Θα ακούσω προσοχή τους συναδέλφους και με τα σχόλιά τους ελπίζω να εκπονήσω ένα πολύ καλύτερο σχέδιο έκθεσης. Ελπίζω αύριο να έρθουν όλοι οι σκιώδη στην ακρόαση. Θέλω να ακούσω τους εκπροσώπους των υπηρεσιών, των οργανισμών, ποια άποψη έχουν, πώς επηρεάζει ο κανονισμός κατά τη γνώμη του τη θέση τους, γιατί υπάρχει ένα νομικό κενό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το καλύπτει μέσα στο παράρτημα ε, της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γνωρίζω όμως ότι δεν συμφωνεί για αυτό το θέμα η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Ε, ε, συμφωνώ με τις ε, παρατηρήσεις σας, κυρίως με αυτή την τελευταία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρέπει να είναι υποδειγματικό σε θέματα διαφάνειας. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι έχουμε μια κουλτούρα διαφάνειας μέσα στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. ιδίας εμπειρίας ξέρω ότι κυρίως το Συμβούλιο είναι ε, εξαιρετικά απρόθυμο να ε, ε, παράσχει πρόσβαση στα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις και στις εξωτερικές του σχέσεις χρησιμοποιεί διάφορες προφάσεις για να κρατά μυστικά τα έγγραφα. θυμηθείτε τι έγινε με το άκτα. Βέβαια δεν του περνάει το Συμβούλιο πάντοτε και όπως και στη ΣΥΠΑ υπάρχει ένα καταπληκτι... ένας καταπληκτικός νόμος για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Ελπίζω να δώσουμε και εμείς το παράδειγμα αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κάσμα ξαναζήτησε το λόγο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, Πρόεδρε. Ήθελα πριν αρχίσουμε τη συζήτηση να διευκρινίσω ότι... Ε, η αναφορά σε αυτό τον Αμερικανικό νόμο για την ελευθερία ενημέρωσης ε, κάναμε τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Καπιτάνη ε, με εκπροσώπους του Καπιτολίου πριν τον κανονισμό Είπαμε ότι αν τα καταφέρναμε και τα καταφέραμε θα ξεπερνούσαμε ε, τα επιτεύγματα αυτού του Αμερικανικού νόμου για την ελευθερία της ενημέρωσης. Ε, βέβαια ε, σε κάποια πράγματα ε, αλλά σε άλλα έχουμε το προβάδισμα στο κομμάτι του κόσμου όπου μένουμε. Νομίζω ότι κάθε προσπάθεια για το ποιος ε, θα είναι ο πρωταθλητής στη διαφάνεια δεν μπορεί παρά να είναι μια καλή προσπάθεια. Έχουν εγγραφεί τέσσερις γκυόμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύσκολο είναι να ξεπεράσει κανείς το Μάικλ Κάσμαν σε αυτό το θέμα, ούτε πρόκειται να αποπειραθώ εγώ κάτι τέτοιο. Είναι μια καταπληκτική βάση για συζήτηση η έκθεσή του. Έχει κάνει πολλές καλές προτάσεις. Πρέπει να σας πω όμως το είπε και ο Μάικλ, ε, όταν συνεδρίασαν οι ηγητές, δεν μπόρεσα να πάω όλο μου, το είπαν οι συνεργάτες μου, ότι και ε, η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η γραμματεία μας δηλαδή, προειδοποίησαν αυστηρά για το τι θα σημαίνει αυτό για το Κοινοβούλιο. Και το λέω αυτό σε εσά, Πρόεδρε. Ε, καλά, αυτό δεν μπορεί να είναι η κουλτούρα και ο πολιτισμός και η στάση του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι θα μπορέσουν να διαρρεύσουν ή να δημοσιεύονται στοιχεία για τα οικονομικά μας. Θα πρέπει εμείς να το χειροκροτούμε αυτό, όχι να το φοβόμαστε. Είμαστε εκπρόσωποι του λαού εδώ και δεν θα πρέπει να έχουμε τίποτα να κρύψουμε ούτε να φοβηθούμε και για την οικονομική μας διαχείριση. Κάτι άλλο που αναφέρει η τροπολογία 32 για τον ορισμό των εγγράφων ίσως να κοιτάξουμε ε, τα θέματα που είναι θέματα προσωπικού ή θέματα ιατρικού απορρίτου, γιατί έχουμε προβλήματα έτσι κι αλλιώς. Γιατί οι υπαλλήλοι μας δίνουν πολλά στοιχεία που είναι και ιατρικά απόρριτα και συγκεντρώνονται αυτά ε, και καλό είναι να δούμε πώς θα τα προφυλάσσουμε για να αποφύγουμε έτσι δύσκολες καταστάσεις και ό,τι άπτεται της ιδιωτικής σφαίρας και της προσωπικής ζωής του καθενός. Αυτό θα πρέπει να παραμένει ως εξαίρεση, αλλά τα υπόλοιπα και τα οικονομικά νομίζω ε, πρέπει να είναι ε, δημόσια. Ε, μερικές ε, έτσι, παρατηρήσεις. τροπολογία 19 για το Μητρό των Ομάδων Πίεσης στο Λόμπι αν είναι υποχρεωτικό να είναι υποχρεωτικό όμως, γιατί αυτό είναι καλό, αλλά η τροπολογία 19 δεν είναι σαφής αν θα είναι υποχρεωτική εγγραφή. Στη συνέχεια, τροπολογία 22 για ενδεχόμενη προσωρινή μη διάθεση ή άνηση διάθεσης ε, των ε, στοιχείων των εγγράφων, το δεδομένο αυτό πώς θα γίνεται. Θα πεις ξαφνικά ότι για μια περίοδο το τάδε έγγραφο δεν είναι διαθέσιμο και μετά θα ξανά είναι. Και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Μετά, ε, κάτι που προτείνεται ε, για μια επιτροπή να ελέγχει ε, ε, τη διαβάθμιση των εγγράφων, αν θα είναι τριμελής ή επταμελής, δεν ξέρω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να εκπροσωπούνται όλες οι ομάδες εκεί στην Επιτροπή αυτή και υπάρχουν και διάφορα συστήματα, ένα σωρό ε, λογιστικά για να μοιράζουμε τις θέσεις. Αλλά ε, πρέπει να τα συζητάμε όλοι και να τα συναποφασίζουμε και είναι δύσκολο να το κάνουμε αν είναι τριμελής και δεν έχουν όλες οι ομάδες ε, εκπροσώπηση. Και στην τροπολογία 50 είναι το κόστος που θα επομιστεί κάποιος που ζητάει πληροφορίες. Ε, εντάξει, έχει και ένα κόστος αυτό, το ξέρουν και οι υπάλληλοι, γιατί όποιο ζητάει μια πληροφορία, καλό είναι να... Ε, επομίζεται αυτό το κόστος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Στο μεταξύ έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Οι επόμενοι εμιλητές παρακαλώ να προσπαθήσετε να είστε πιο σύντομοι. Κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για τη διαδικασία και την πιο πρόσφατη της έκθεσης. Ε, όταν συνεδρίασαν οι σκιώδεις ηγητές παρακάλεσα η συζήτηση για την έκθεση να αναβληθεί μέχρι να έχουμε τις μεταφράσεις στις διάφορες γλώσσες μας. Είχε την καλοσύνη να το δεχτεί ο εισηγητής. Έχουμε το δικαίωμα να εργαζόμαστε και στη μητρική μας γλώσσα εδώ μέσα. Και πρέπει να σας πω ότι η γερμανική μετάφραση έφτασε την Παρασκευή στις 12 η ώρα, παραμονές Σαββατοκύριακο, και οι άλλες γλώσσες στις 7 το απόγευμα. Και πρέπει, λέει, να προετοιμαστείς μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ε, γρίφος για μένα. 11 χρόνια είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η Επιτροπή μας είναι από τις λίγες επιτροπές όπου ε, υποχρεωνόμαστε πολύ συχνά να εργαζόμαστε σε ξένες γλώσσες. Εγώ μπορώ να δουλέψω και στα αγγλικά, αλλά δεν το θέλω. Και είναι πολύ ευαίσθητα και λεπτά τα ζητήματα αυτά και θα πρέπει να μπορεί ο καθένας να δουλεύει στη μητρική του γλώσσα. Θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό και θα το ξαναπώ στην Επιτροπή μας. Τώρα, έρχομαι στην έκθεση την ίδια, στο σχέδιο. Τα γενικά προβλήματα που είχα μέχρι τώρα δεν έχουν ε, λυθεί ακόμα όλα, το ξέρει και ο εισηγητής αυτό. Ε, κατά την άποψή μου δεν έχουν διευκρινιστεί πολλά πράγματα και δεν έχουν ε, ε, περιχαρακωθεί. Για παράδειγμα, τι είναι έγγραφο, δεν ξέρουμε καν τι είναι έγγραφο, ο ορισμός του εγγράφου. Θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρος. Και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα έγγραφο και μια πληροφορία. Υπάρχει διαφορά. Αν ανοίγω εγώ την πρόσβαση σε έγγραφα και είναι δημόσια ή αν είναι δημόσια μια πληροφορία η πληροφόρηση να είναι διαθέσιμη. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά. Μετά, θα πρέπει να γίνει ένας αφέστατος διαχωρισμός, η πρόσβαση του κοινού σε εμπιστευτικά έγγραφα και στις διοργανικές συμφωνίες για την πρόσβαση των θεσμικών οργάνων σε εμπιστευτικά ή απόρριτα έγγραφα και όχι του κοινού. Έχω λίγο την εντύπωση ότι προσπαθεί ο εισηγητής έτσι να έχει συνολική πρόσβαση μέσω των ε, διοργανικών συμφωνιών. Και κάπως να τις τροποποιήσει αυτές τις συμφωνίες μέσω της έκθεσής του. Δεν νομίζω ότι είναι δική μας δουλειά αυτή, στην έκθεση αυτή. Εδώ μιλάμε για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Κάτι άλλο που θα πρέπει να λυθεί για μένα και να διευκρινιστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα πώς συμμετέχει σε αυτό και ε, ως θεσμικό όργανο ή ως ε, νομοθέτης διότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο γιατί αυτό εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διαφορετικά έγγραφα, σε διαφορετικού τύπου έγγραφα. Για πάλι δεν το έχω καταλάβει τελείως. Άλλο θέμα τώρα. Η πρόσβαση στα έγγραφα για μέλη του Κοινοβουλίου, για τους συνεργάτες, βοηθούς, υπαλλήλους και για την κοινή γνώμη. Και πάλι αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και από αυτό που λένε οι συνάδελφοι δεν έχω καταλάβει, έχω μπερδευτεί περισσότερο. Εντάξει, λένε ότι όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων και των βουλευτών δεν θα πρέπει να είναι δημόσια. Προφανώ υπάρχει και εδώ προστασία δεδομένων. Από την άλλη λέει ο εισηγητή ότι. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Για ακούστε, συνάδελφοι. Για τους βοηθούς, ας πούμε, και μόνο, θα πρέπει να είναι όλα δημόσια και διερωτώ με. Η προστασία δεδομένων δεν ισχύει ξαφνικά για τους βοηθούς μας. Στη Γερμανία, που υπάρχει το φορολογικό απόρριτο και δεν μπορεί ο καθένας να δημοσιεύει ας πούμε και τα ιατρικά του δεδομένα. Υπάρχει και το ιατρικό απόρριτο. Υπάρχουν στοιχεία που άπτονται της προσωπικότητας του ανθρώπου και δεν μπορούν να είναι δημόσια. Επειδή είναι υπάλληλοι του κοινοβουλίου, δηλαδή πρέπει να είναι διαφανείς. Και αυτό πάλι δεν το έχω καταλάβει. Και τι είναι το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Γιατί αυτό λέει ο εισηγητής, εφόσον υπάρχει ένα ε, υπέρτατο συμφέρον που το επιτάσσει και τα λοιπά, θα πρέπει αυτό να επιτρέπεται. Και ποιος το ορίζει αυτό αν υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον. Και αυτό θέλει ορισμό. Γιατί να προέχει το δημόσιο συμφέρον και πότε προέχει. Είναι θέμα ερμηνεία κατά το δοκούν όποιο το αποφασίζει αυτό. Για κοιτάξτε το και αυτό σα παρακαλώ. Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι σε πολλού τομεί για να ξέρει ο καθένα μετά ποιο έχει πρόσβαση σε ποιε πληροφορίε και να κανονίζει την πορεία του. Ένα πρώτο τελευταίο, γιατί έχω κι άλλο. Ε, πώς μπαίνει εδώ ο διαμεσολαβητή στη λήψη των αποφάσεων για τη δημοσίευση ή τη μη δημοσίευση κάποιων εγγράφων. Και πάλι ανησυχώ ότι αυτό υπερβαίνει την εντολή του διαμεσολαβητή. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό ως ρόλο. Μήπως να αλλάξουμε την εντολή του. Το θέλουμε. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο διαμεσολαβητής. Ένα πρόσωπο να ε, αναλαμβάνει την ευθύνη να παίρνει αυτή την απόφαση. Και το τελευταίο, επί της ουσίας πάντα, στόχος αυτού του κανονισμού πιστεύω πρέπει να είναι να ενημερώνονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι σε θέση να παρακολουθούν πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στα θεσμικά όργανα. Μάλιστα, όλοι το επιθυμούμε αυτό, να είναι διάφανη η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην θεωρούν οι πολίτες ότι αποκλείονται ή ότι τους ποδηγετούμε ή τους χειραγωγούμε. Όλα αυτά καλά, αλλά εάν δεν προσέξουμε, ο κανονισμός αυτός, τουλάχιστον όπως έχει τώρα η έκθεσή σας και το σχέδιο, θα επιφέρει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιθυμούμε. Δηλαδή, θα τον κατακλείσουμε τον πολίτη με όλες αυτές τις πληροφορίες. Μια πλημμύρα και οι από τις πληροφορίες αυτές είναι και τελείως άχρηστες. Γιατί είναι σε μια διαδικασία που βρίσκεται στην πορεία και ο πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι είναι αποφασιστική σημασία έγγραφο ή όχι όταν τον κατακλείσεις με μια ε, πληθώρα εγγράφων. Δεν μπορεί να διακρίνει το σημαντικό και το επουσιώδης. Και αυτό θα κάνει την Ευρώπη ακόμα πιο θολή για το μέσο πολίτη. Και τέλος μια ερώτηση. Ε, η πρόεδρος, μήπως να συντομεύατε, κυρία Σόμερ. Ναι. Η Επιτροπή Αναφορών ανέβαλε την ημερομηνία για τη γνωμοδότησή της και μπορεί να τη φέρει και μετά το καλοκαίρι. Να υποθέσω λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης αλλάζει αντίστοιχα και θα προσανατολιστούμε στην Επιτροπή Αναφορά. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που σας διακόπτω, αλλά έχω πάρα πολλούς ομιλητές και αν ο καθένας ομιλεί τόσο πολύ δεν προλαβαίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, αλλά προσπαθήστε να είστε όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται. Πρόντς. Προφανώς και είμαι υπέρ της πρόσβασης στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα αυτό όμως όταν είναι γραμμένο σε περίεργες, με περίεργο τρόπο και σε περίεργες γλώσσες δεν γίνεται κατανοητό. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει έστω και ένας πολίτης καλλιεργημένος και έξυπνος ο οποίος θα κατανοήσει το έγγραφο αν τυχόν δεν έχει προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Ακόμα και στη δική μου γλώσσα τα έγγραφα όταν τα διαβάζω ε, πραγματικά είναι σαν να έχουν ε, μεταφραστεί ε, σε κάποιες γλώσσες οι οποίες πλέον είναι νεκρές εδώ και αιώνες, είναι πλήρως ακατανόητες και γι' αυτό δημιουργείται μια νομική αβεβαιότητα και υπάρχει μια έλλειψη κατανόησης αυτών των συγκεκριμένων εγγράφων. Εγώ δεν είμαι γενικά υπέρ της ευρωπαϊκής πρακτικής, αλλά καλό θα ήταν να υπήρχε και μια εταιρεία η οποία να ελέγχει τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε όταν γράφουμε επίσημα κείμενα. θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω την αντίληψη του Κάσμαν. Αν συγκρίνει κανείς την αρχική πρόταση της Επιτροπής και μετά το κείμενο που προτείνει ο Κάσμαν, είναι σαφές ότι είναι πληρέστερο και οι προτάσεις της Επιτροπής δεν εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους δίδει η συνθήκη της Λισαβόνας. Λοιπόν, διαφάνεια, προσβασιμότητα και δεν μιλάμε μόνο για φυσική προσβασιμότητα, αλλά ακριβώς και επίπεδο δυνατότητας κατανόησης των εγγράφων αυτών πρέπει να είναι γραμμένα με τρόπο έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά. Η διαπραγμάτευση δεν είναι εύκολη αλλά θα πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να είναι πρωταθλητής θα έλεγα το Κοινοβούλιο στην προσπάθεια για μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολότερη κατανόηση. Ευχαριστώ κύριος Γιακολίνο. Είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ξεκινήσω από την υπόθεση τροποποίησης του κανονισμού του 2001 εξέτασα με αρκετή προσοχή τα κείμενα και άκουσα προσεκτικά και αυτά τα οποία υπόθηκαν σε αυτήν την αίθουσα. Ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος και οι στόχοι τους οποίους έχει και ο κύριος Κάσμαν είναι πλήρως κατανοητοί μεγαλύτερη πρόσβαση, καλύτερη κατανόηση, ουσιαστικά δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία, δηλαδή λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι σε θέση να ελέγχουν με σωστό τρόπο τους εκπροσώπους τους. Διάβασα επίσης ε, προσεκτικά και την ονοματολογία των νομικών πράξεων ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς τις διαφορές ανάμεσα σε νόμους, κανονισμούς, ε, οδηγίες κτλ. Πάντως, μία πρόταση σαν αυτή την οποία κάνει ο κύριος Κάσμαν και το ξέρει ο κύριος Κάσμαν έχει ένα κόστος. Ένα κόστος το οποίο δεν είναι ασήμαντο θα έλεγα. Σήμερα αγαπητέ κύριε Κάσμαν ψηφίσαμε καταρχάς Ξέρετε, πήραμε την απόφαση τη συγκεκριμένη για την διακυβέρνηση του ε, διαδικτύου έτσι ώστε να υπάρξουν μεταφράσεις και σε άλλες γλώσσες εκτός αγγλικής όπως τα Ιταλικά κτλ. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να μην αγνοήσουμε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο οργάνωσης των εργασιών μας. Αν θέλουμε ένα τόσο υψηλό επίπεδο πρόσβασης τότε θα πρέπει να καλύψουμε το νέο αυτό οργανωτικό πρότυπο το οποίο θα κοστίσει πολύ. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές δεν αξίζει να δημοσιεύονται όλα σε όλες τις γλώσσες. Σαν παράδειγμα η επίσημη δημοσίευση των προπαρασκευαστικών πράξεων Εκεί θα μπορούσαμε να τα μεταφέρουμε αυτά σε όλες τις γλώσσες φυσικά και προς ανάγνωση από όλους με συνοπτικό τρόπο να παρουσιάσουμε συνόψεις, να παρουσιάσουμε ε, κάποιες περιλήψεις όπου αυτό φυσικά είναι ε, αποδεκτό. Εν μία τελευταία παρατήρηση εδώ μερικές φορές μια πολύ ελεύθερη πρόσβαση, όσο δίκαιη και αν είναι, μπορεί να δημιουργεί ε, κάποιες θα έλεγα μορφές περιέργειας οι οποίες ε, δεν είναι πάντα θεμητές. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Προτελευταίος ο μιλητής Αλφάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κάσμαν. Ξέρω ότι ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με τα θέματα της διαφάνειας και προσπαθεί έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν όλο περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στις ε, εργασίες μας. Πράγματι θα πρέπει το κοινό να έχει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα που αφορούν θέματα όπως το PNR, τα SWIFT κτλ. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Κάσμαν γιατί ίσως να μην έχω καταλάβει κάποια πράγματα καλά. Υπάρχει το άρθρο 33 της παραγράφου 9 το οποίο λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα μόνο μέσω συγκεκριμένων εγκεκριμένων ομάδων βουλευτών. Θα ήθελα εδώ να με βοηθήσετε να καταλάβω. Ο περιορισμός αυτός ε, είναι ένας περιορισμός όπως λέει η λέξη. Μπορεί να ξεπεραστεί με κάποιο τρόπο για να υπάρξει σωστότερη ενημέρωση. Ε, επίσης ε, ένα άλλο άρθρο σας αναφέρεται στις δυνατότητες ε, να εφεσιβάλει κανείς την ε, δυνατότητα ή μη δυνατότητα πρόσβασης σε, συγκεκριμένες, ε, σε συγκεκριμένα κείμενα και έγγραφα. Θα ήθελα να μου δώσει κάποιες εξηγήσεις, να καταλάβω επίσης γιατί ο κύριος Κάσμαν τροποποιεί το άρθρο 39 το οποίο είχε γίνει ήδη στο παρελθόν δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μία τελευταία παρατήρηση είναι να μας πει ποια είναι τα τμήματα του παλαιότερου κανονισμού τα οποία χωρίς τροπολόγηση μπορούν να περάσουν και να ισχύσουν άμεσα στον καινούριο. Στο μεταξύ έχουμε άλλον έναν ομιλητή στον κατάλογο, αλλά πραγματικά τώρα ε, η, κυρία, η κυρία Βέιμπερ και ο κύριος Μάλκοβερ θα είναι οι τελευταίοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Εδώ και καιρό προσπαθούμε να ρυθμίσουμε το θέμα της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα με αυτόν τον κανονισμό και τι να σας πω ξαφνιάζομαι που εξακολουθούν να υπάρχουν σχόλια που δεν αποσκοπούν στην αναβάθμιση του κειμένου, αλλά αποσκοπούν στο να εκδηλώσουμε μια προθυμία γιατί χρειαζόμαστε τη ρύθμιση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πώ ακριβώς, τι μήνυμα θα περάσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Πώς μπορούμε να μιλάμε για το έλλειμμα, το δημοκρατικό έλλειμμα, ε, ε, για την απόσταση που χωρίζει την Ένωση από τους πολίτε της και ταυτόχρονα να μην μπορούμε να κάνουμε έναν πλήρη κανονισμό για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οφείλω να πω ότι την τελευταία δεκαετία σε χώρες που δεν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω και ως δημοκρατικές υπάρχει νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και βλέπω να μην υπάρχει τέτοια νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα είναι ντροπή. Ε, πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στους πολίτες μας. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία και με επικοδομητικό τρόπο και να μην ε, υποβάλουμε τόσες πολλές τροπολογίες ώστε να αποδυναμώσουμε το κείμενο γιατί δεν πρέπει να είναι αυτός ο στόχος μας. Όλοι γνωρίζουμε δε πως ε, πίσω από αυτή την εμπιστευτικότητα, πίσω από την απροθυμία που υπάρχει για την πρόσβαση, ε, δίκιο δεν έχουν οι πολίτες να υποπτεύονται διαπλοκή και διαφθορά υπάρχουν πράγματα που δεν είναι σαφή ή μπορεί να δώσουμε την εντύπωση ότι η καρφάκι δεν μας καίγεται για τους πολίτες. Μας ψηφίζουν αλλά μετά δεν θέλουμε να είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις μας. Ε, και όταν πρόκειται για αναθεώρηση και εξέταση των πράξεών μας λέμε όχι ε, δεν έχετε καμία δουλειά να βλέπετε τα έγγραφα, δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μακόβη, ε, θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω ε, την αρχή πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι ε, ενίοτε είναι υπερβολικός ο όγκος των πληροφοριών ή ότι είναι πληροφορίες που δεν είναι χρήσιμες στους πολίτες. Μα δεν θα αποφασίσουμε αυτό. Εκείνοι θα αποφασίσουν. Θα διαλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και θα αποφασίσουν αν τους ενδιαφέρουν ή όχι. Δεν αποφασίσουμε εμείς αν πρέπει να παράσχουμε στο κοινό ενημέρωση και πληροφορία. Ε, τώρα το ότι δεν είναι βανάγνωστα τα κείμενα αυτό είναι πρόβλημά μας ε, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιορίζουμε την πρόσβαση στα έγγραφα επειδή είναι περίπλοκα, ε, ε, έχουν κακή διατύπωση τα κείμενα και είναι δυσανάγνωστα. Οφείλουμε να έχουμε καλή επικοινωνία με το κοινό, να κατοχυρώνουμε την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Αυτό είναι δικό μας καθήκον, είναι πρόβλημα που εμείς πρέπει να λύσουμε. Δεν είναι επιχειρήματα όλα αυτά που ακούσαμε, επιχειρήματα μπορούμε να προτάξουμε για να περιορίσουμε την πρόσβαση του κοινού. Είναι προβλήματα που πρέπει να λύσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Μακόβη. Πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν συντομία και κατόπιν στον εισηγητή, να κάνω κι εγώ κάποιε παρατηρήσει. Πρώτον, υπάρχει σαφή αντίθεση ανάμεσα ε, στον βαθμό διάβρωση τη ιδιωτικότητα των πολιτών τα τελευταία δέκα χρόνια προβάλλοντα το επιχείρημα ότι αν δεν έχετε τίποτα να κρύψετε δεν έχετε και τίποτα να φοβηθείτε. Ε, οι δημοσίες αρχές ε, πρέπει να έχουν πρόσβαση όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αλλά αν αντιστρέψετε αυτή τη λογική και την εφαρμόσετε και σε εμά ε, στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, ε, τα εθνικά θεσμικά όργανα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, ε, τι να έχουν, θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερα προτερήματα και κρύβουν τις πληροφορίες. Άρα υπάρχει ανισορροπία. Δεύτερον, Μάικλ, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξή. Είπε ότι το μέσο που αναμένεται να εγκριθεί θα είναι ισχυρότερο και από τον Αμερικανικό νόμο για την ελευθερία της πληροφόρησης. Δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι πεπισμένη ότι με αυτή τη νομική πράξη θα έχουν ένα ισχυρό εργαλείο οι πολίτε στα χέρια του. Το θέμα ποιο είναι ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να κρύβονται πάντοτε πίσω από το επιχείρημα τη επικουρικότητα ή των διεθνών σχέσεων. Πάντοτε βρίσκουν ένα λόγο, μία πρόφαση να πούν ότι βεβαίω θα θέλαμε να σα κοινοποιήσουμε, να δημοσιεύσουμε το έγγραφο, γιατί, αλλά δεν μπορούμε γιατί δεν θέλουν οι εταίροι μα ή δεν θέλουν τα κράτη-μέλη. Και έχω δει πολλαπλά τέτοια παραδείγματα για του σαρωτέ σώματο, παραδείγματο χάρη. Πήραμε πολλές πληροφορίες από τους Αμερικανούς φίλους μας που τις είχαν ε, ε, βρει ε, μέσω ερωτηματολογίων για τις προδιαγραφές, τεχνικές προδιαγραφές των σαρωτών και όταν εμείς ζητήσαμε αντίστοιχες πληροφορίες από τις δικές μας εθνικές αρχές δεν τις λάβαμε. Τις πήραμε από τους Αμερικανούς, τις είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες τις ζητήσαμε και από τις εθνικές αρχές, πλην όμως δεν τις λάβαμε. Και δεν υπήρχε καμία ευρωπαϊκή αρμόδια αρχή στην οποία θα μπορούσαμε να αποταθούμε για να τι αποκτήσουμε τι πληροφορίε. Υπάρχει νομικό κενό, υπάρχει μια έλλειψη λόγω της οποίας ε, για να δούμε τι κάνουν οι κυβερνήσεις μας και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθυνόμαστε στους Αμερικανούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ να είστε πραγματικά σύντομοι. Δεν έχουμε ακόμη καθυστερήσει, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Τρία λεπτά κατά ανώτατο όριο για να ακούσουμε και πάλι τον εισηγητή μετά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Συγχαρητήρια στον κύριο Κάσμαν που επανέφερε στην επικαιρότητα το θέμα και ξεκίνησε εκ νέου συζήτηση. Υποστηρίζουμε τη συζήτηση αυτή και θέλουμε να υπάρξει επικοδομητικός διάλογος. Αφορά ο κανονισμός αυτός τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι το θέμα και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, το κέντρο της προσπάθειάς μας, το κέντρο τη της προσοχής θα έλεγα του νομοθέτη πρέπει να είναι τα δικαιώματα των πολιτών πρόσβαση στις εργασίες των θεσμικών οργάνων. Παράλληλα λοιπόν με τις συζητήσεις που γίνονται ε, σε διοργανικό επίπεδο για τις δυνατότητες θεσμικής πλέον ή οργανικής πρόσβασης του ενός οργάνου στα έγγραφα του άλλου, δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα εδώ νομικών δικαιωμάτων που εδράζονται στη συνθήκη γύρω από τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες όχι στην παραγωγή νέων μορφών ενημέρωσης ή πληροφορίας, αλλά στα έγγραφα και στις εργασίες των οργάνων. Νομίζω ότι όλοι το επιθυμούν αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που κάτι τέτοιο δεν το επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την προσπάθεια αυτή και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την νομολογία η οποία έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Έχουν υπάρξει σε ορισμένους τομείς ορισμένες αμφιβολίες και χρειάστηκε το δικαστήριο πλέον να πάρει την απόφαση του να διαιτητεύσει και να αποφασίσει. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει σε πολιτικό επίπεδο να παίρνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, νομίζω ότι γνωρίζει ότι πρέπει να εξισορροπήσει πρώτα τον κανονισμό για την πρόσβαση στα δεδομένα ε, με τα δικαιώματα ε, των πολιτών Ξέρετε ότι οι δημόσιοι μηχανισμοί για διάφορους λόγους σε εθνικό επίπεδο συγκεντρώνουν τεράστιες ποσότητες στοιχείων και δεδομένων για διάφορους λόγους ε, ασφαλείας κτλ. Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν ε, ε, στοιχεία ιδιωτικά, να μην χρησιμοποιούνται και έτσι λοιπόν ο 1049 και ο 45 θα πρέπει από κοινού να επιδιωχθεί να βελτιωθούν. Θα ήθελα να εμείνουμε λίγο στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σε ορισμένες προτάσεις τις οποίες θεωρεί πολύ σημαντικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απλά ο διαχειριστής, αν θέλετε, των πολιτικών αυτών. Είμαστε και πολιτικό σώμα και έχουμε το δικαίωμα της πολιτικής πρωτοβουλίας και έχουμε ένα επιπλέον ακόμα ρόλο για τον οποίο ανησυχούμε. Τελειώνω εδώ, είναι το τελευταίο μου σημείο Είμαστε η υπηρεσία η αρμόδια για τον ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι θέλουμε να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ρόλο αυτό, έναν ρόλο ο οποίος ασκήθηκε αποτελεσματικά προς όφελον όλων των ενδιαφερομένων. Εννοείται λοιπόν ότι τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα οποία έχουμε πάρει με εισαγγελική βοήθεια στις 5 η ώρα το πρωί μετά από εισβολές σε εισαγωγικά σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, προφανώς αυτά δεν μπορούμε να τα δημοσιεύουμε εύκολα και να τα ανοίξουμε σε όλους τους ενδιαφερομένους με καλό στόχο πιθανώς. Αυτό ελπίζω να το καταλάβετε. Κύριε Κάσμαν, θέλετε να κλείσετε σε λίγα λεπτά τη συζήτηση θα μπορούσα, αλλά θα με κατηγορήσετε ότι δεν έχω απαντήσει σε όλα τα ε, ερωτήματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ όλους όσους ε, έχουν συνεισφέρει στη συζήτηση, ακόμα και αυτούς που διαφωνούν με αυτά τα οποία είπα. Οι τροπολογίες 32, η τροπολογία 32, συγγνώμη, Πράγματι θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος, μια λίστα εδώ. Αλλά θα πρέπει όμως να δούμε ποια θα είναι η νομική βάση για την οποία ή πάνω στην οποία θα βασίζεται ακριβώς αυτή η υποχρεωτική εγγραφή. Η κοινότητα δεν είναι αυγό έτσι ώστε να το φάει κανείς μελάτο ή ομελέτα. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε εκ των προτέρων για τη φύση των εγγράφων αυτών. Το λέω σε όλους τους συναδέλφους και πρέπει να το καταλάβουμε. Οι φιλοδοξίες μου δεν είναι ο χαμηλότερος δυνατός παρανομαστής. Μη γελιέστε. Ζητώ και ακριβώς το ίδιο περιμένω και από όλους ε, τους βουλευτές να θεωρήσουν ε, ότι ε, ο κανονισμός 46 του 2000 σαν παράδειγμα είναι εξαιρετικά σημαντικός Δημιουργείται λοιπόν ένας πανικός κυρία Σόμερ, ο οποίος προέρχεται και από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από ε, εκπροσώπους γενικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα τι σύγχυση είναι αυτή. Εδώ αναφερόμαστε ε, ε, στην δυνατότητα ε, φυσικά και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα άλλων οργάνων, αλλά μέσω των διοργανικών συμφωνιών. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Ήδη από το 2001 είχαμε τον πρώτο κανονισμό για την πρόσβαση στα έγγραφα ανάμεσα στα μεγάλα θεσμικά όργανα. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όταν πάει καλά πρέπει να το αφήσουμε όπως είναι και όταν κάτι δεν πάει καλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε εισαγωγικά να το επισκευάσουμε. Λοιπόν, ακούμε να ανησυχούν διάφοροι δικηγόροι, ε, λόμπιστ, θα πρέπει όμως ε, να φανούμε ρεαλιστές και εδώ έρχονται και οι Αμερικάνοι. Λέγουν ότι όταν εσείς στην Ευρώπη αν έχετε έναν δημόσιο κατάλογο εγγραφή σαν παράδειγμα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Εμείς κάτι τέτοιο δεν το έχουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Για την κυρία Σόμερ οι μεταφράσεις οι οποίες είναι διαθέσιμος ε, την τελευταία στιγμή μόνο. Ναι, πράγματι, την Παρασκευή μας ήρθαν οι μεταφράσεις, γιατί να μην δουλέψω και το Σαββατοκύριακο. Ήρθα από ταξίδι, παρόλα αυτά δούλεψα το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό είμαστε εδώ. και πράγματι οι αρχές επί του προϋπολογισμού θα πρέπει να μας δώσουμε περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να έχουμε τις πληροφορίες όλες αυτές τις γλώσσες μας για να μπορέσουμε πολιτικά να είμαστε ισότιμα όλοι με τον ίδιο τρόπο αποτελεσματικοί. Βέβαια υπάρχουν κάποια θέματα πάνω στα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε, το αναγνωρίζω αυτό για την κυρία Μακοβέη σαν παράδειγμα. Η φήμη σας κυρία Μακοβέη υπέρ της ε, ε, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα σας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χαιρετήσουμε σαν ένα εξαιρετικό παράδειγμα προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη αλλά δεν πρέπει όμως να φανούμε πατερναλιστικοί και να πούμε ότι μα είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που δεν έχει νόημα να τους τα δώσουμε όλα αυτά δεν τα δίνουμε μόνο στον μεμονωμένο πολίτη, τα δίνουμε σε δικηγόρους, σε νομικούς, σε δημοσιογράφους, ενημερώνουμε όσους θέλουν να ενημερωθούν. Συνεπώς λοιπόν το επιχείρημα αυτό δεν είναι σωστό. Οι προθεσμίες. Κοιτάξτε, ε, όσο περισσότερο μεγαλύτερο είναι το χρονοϊκό διάστημα διάθεσης, ε, τόσο το καλύτερο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το επιχείρημα αυτό για να περιορίζουμε την πρόσβαση. Προφανώς, αν υπάρχει σαν παράδειγμα μια θαλάσσια μόλυνση και κάποιος ζητάει πληροφορίες και θέλει να μάθει τι στοιχεία έδωσε η BP σαν παράδειγμα, προφανώς θα πρέπει να είμαστε σε θέση κάποια από τα στοιχεία αυτά να καλύψουμε με τα στοιχεία αυτά, να καλύψουμε τις ανάγκες τις οποίες έχει το κοινό και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κύριε Μπρόντς, ίσως να μην είναι άποψη του κόμματός σας. Αν θέλετε να το διατυπώσω καλύτερα, βοηθήστε τα Κίνγκα Πράγματι θα υπάρξουν ε, δύσκολες διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι δεν θα ε, κρατήσουν όμως πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι διαπραγματεύσεις αυτές. Είμαι ε, βέβαιος ότι θα κατηγορηθώ ότι δεν ακολουθώ σε ορισμένες περιπτώσεις ε, τον σωστό δρόμο. Πάντως αυτό το οποίο ε, είναι σαφές είναι ότι θα πρέπει ο πολίτης ο οποίος πληρώνει να καλύπτει τις προσδοκίες του. Η αναφορά που γίνεται σε κάποιες προσωρινές διαδικασίες ε, οι οποίες δεν είναι απόλυτα ανοιχτές και δεκτικές σε έλεγχο του κοινού εδώ έρχεται το θέμα της επιμέρους πρόσβασης που μπορεί να ακολουθήσει ετεροχρονισμένα σαν παράδειγμα για λόγους πρακτικούς βέβαια. Είναι κάτι το οποίο όμως η συνθήκη της Λισαβόνας δεν δέχεται εύκολα αν θέλετε γιατί θέλει οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχουν στην διαδικασία και αν έρχονται εκ των υστέρων στη διαδικασία δεν το πετυχαίνουν αυτό. Ε, τέλος υπάρχει το θέμα αυτής της Επιτροπής, της ομάδας των βουλευτών που είναι 7 ή λιγότεροι περισσότεροι. Εδώ το θέμα είναι προσυζήτηση. Για την τροπολογία 30 αφορά πάντα την πρόσβαση των βουλευτών στα έγγραφα. Αυτά τα οποία προτείνω να απορριφθούν αφορούν το καθεστώς των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκανα κάποιες αλλαγές έτσι ώστε το ΕΛΚ να μας υποστηρίξει αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά δεν ε, υποστήριξαν τις προτάσεις που είχα κάνει. Ε, εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε εμείς εδώ κάποιες προτάσεις ή τροπολογίες οι οποίες να αλλοιώνουν ή να ενισχύουν το καθεστώς του βουλευτού κτλ. Υπάρχει αναφορά και σε αυτά τα οποία είπατε και πολύ σωστά στο δημοκρατικό έλλειμμα και αν δεν ασχοληθούμε με την κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος ότι ουσιαστικά θα ενθαρρύνουμε τη μεγέθυνσή του. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά πάλι και την κυρία Μακοβέη. Το κοινό είναι αυτό που θα αποφασίζει τι θέλει. Εμείς θα θέσουμε στη διάθεση του κοινού τους μηχανισμούς για να πετυχαίνει τον στόχο αυτό με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο το βέτο της τρίτης πλευράς, από άλλες χώρες δηλαδή. Πράγματι προσπαθήσαμε να το λύσουμε σαν Επιτροπή, σαν Συμφούλιο, σαν Κοινοβούλιο και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν τα πετύχαμε μέχρι τώρα τα πράγματα όπως τα θέλαμε. Σύμφωνο και με τον Γένσε ότι είπε, αλλά τα θέματα του ανταγωνισμού καλύπτονται ε, αυτή τη στιγμή ε, και από νομοθετικές ρυθμίσεις εφόσον υπάρχει μια έρευνα, μια ανάκριση. Όταν η πληροφορία καθίστεται ε, διαθέσιμη, τότε μπορεί να φανεί ότι μια επιχείρηση ε, που ήταν τμήμα του καρτέλ έδωσε πληροφορίες για να σπάσει το συγκεκριμένο καρτέλ και ε, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα αντικίνητρο για άλλες εταιρείες στο μέλλον. Λοιπόν, είπα ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το οποίο προτείνουν, ελπίζω να το καταλάβετε όλοι, στην ουσία χρησιμοποιούν δυσανάλογα θα έλεγα δυνατές μορφές παρέμβασης για να λύσουν τα προβλήματα τα οποία είναι ελεγχόμενα σε μέγεθος και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή ένα επιπλέον νομοθετικό πλαίσιο. Το θέμα που πρέπει να προωθήσουμε είναι να διοργανώσουμε έτσι τη συζήτηση έτσι ώστε να υπάρξει συζήτηση και η τρίτη πλευρά, ο τρίτος εμπλεκόμενος να έχει πάντα τη δυνατότητα να κρατήσει εκτός διάθεσης κάποια στοιχεία ή κάποια έγγραφα που τον αφορούν και τον φύγουν άμεσα. Να τελειώσω με κάτι το οποίο για μένα είναι σημαντικό, γιατί είμαι εδώ 11 χρόνια, κάποιοι από εσά με ξέρετε. Όταν εμένω σε μία αρχή, το κάνω αυτό ε, όχι για λόγους μαρξιστικούς Α, ή τουλάχιστον με τον Καρλ Μάρξ μπορώ να συμφωνώ, αλλά με τον Γκρούτσο Μάρξ δεν συμφωνώ, που έλεγε ότι αυτή είναι η αρχή στην οποία πιστεύω και αν δεν σας αρέσει θα την αλλάξω. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Νομίζω ότι ακριβώς με βάση την αρχή αυτή στην οποία εμένω κινδυνεύω μερικές φορές αυτά τα οποία προτείνω να μην γίνουν δεκτά αλλά παρόλα αυτά η μάχη η οποία θα δώσω έχει μεγάλη σημασία και αν αποτύχω εγώ θα το αναλάβει άλλος και ε, νομίζω ότι τα θέματα της διαφάνειας και της δεκτικότητας δεν θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα και όλοι θα θέλουν να μάθουν γιατί οι βουλευτές από όλα τα κόμματα μερικές φορές δεν δέχονται να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους, ακόμα και αυτούς με τους οποίους όπως είπα διαφωνώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι ζητάτε το λόγο, αλλά τελειώσαμε, δεν θα δώσω άλλο. Κοιτάξτε λίγο, είναι 5 και 5 η ώρα για να καταλάβετε. Τώρα θα ζητήσουμε το PNR ε, και είμαι ε, εισηγητρία. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα σα είπα ότι πρέπει να φύγω στι 5.30. 25 λεπτά λοιπόν για να συζητήσουμε ε, τις καταστάσεις επιβατών. Θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά σε αυτή τη συζήτηση παρακαλώ να είστε όλοι πολύ πιο σύντομοι. Ζητώ συγγνώμη, έγινε η συζήτηση, τελείωσε. Θα επανέλθουμε σίγουρα σε αυτό το θέμα, είμαι βέβαιη. Η κυρία Γιακοβέη κάτι λέει. Μα θα το ξανασυζητήσουμε, σα είπα. Και τροπολογίε μέχρι τι 10 Ιουνίου πρέπει να κάνετε. Α, no deadline. Εδώ λέει 10 Ιουνίου και τώρα μου λένε ότι είναι ανοιχτή ε, ακόμα η προθεσμία. Ορίστε, κύριε Κάσμαν. Πρέπει να σα πω ότι η κυρία Μακοβέη συμφωνεί μαζί μου και εγώ μίλησα για την προηγούμενη θητεία όταν ψηφίσαμε για τον κανονισμό αυτό. Όχι για σας. Όταν δεν ψήφισε το ΕΛΚ μαζί μου, δεν με υπερψήφισε. Εδώ στην Επιτροπή αναγνωρίζω απολύτω ότι έχουμε σύμπτωση και απόλυτη αιμοφωνία σε αυτό, με, τουλάχιστον με την προσέγγισή μου. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη, θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Θέλω να περάσω στο επόμενο, σας παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι είναι σαφή συζήτηση. Seconds, five seconds. So I said I Πέντε δεύτερα. Είπα ότι δεν συμφωνώ με επιχειρήματα τύπου υπερβολική ε, πληροφόρηση ή περισσότερο ή λιγότερο σχετική πληροφόρηση. Όλα ανοιχτά στο κοινό και το κοινό θα αποφασίσει τι χρειάζεται και τι θέλει να μαθαίνει. Ωραία. Σαφέσταν αυτό. Πάμε παρακάτω. PNR. Ως εισηγήτρια και πρόεδρος σας παρακαλώ, σας ζητώ να συνεργαστείτε και να περιορίσετε τα σχόλιά σας ε, όσο μπορείτε, χωρίς επικαλύψεις και χωρίς επαναλήψεις. Γιατί μπήκε ξανά στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα και δεν το γράφει η ημερήσια διάταξη. Από την περασμένη συνεδρίαση και συζήτηση που είχαμε, πήραμε κοινή αναθεώρηση τη Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Είχατε την ευκαιρία να τη διαβάσετε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ήδη. Και θα πρότεινα το εξή. Να αρχίσει πρώτα η συζήτηση και να κάνετε όλοι τις ερωτήσεις σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ μετά θα τη ζητήσω να απαντήσει. Μερικές ε, ερωτήσεις έχω και εγώ να κάνω. Τις έχουμε στείλει γραπτό στην Επιτροπή. Επανειλημμένος, χωρίς ακόμα σαφή απάντηση. Λοιπόν, θα αρχίσω εγώ, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη και θα ήθελα να κάνετε και σύντομα σχόλια και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινή ενθεώρηση και να ακούσω και τα σχόλιά τους. Γιατί δεν μπορούν να αποκαλύψουν όλες τις προφορίες που έχουν στα χέρια τους ή έχουν πρόσβαση. Γιατί. Και αυτό τι αξία δίνει στην κοινή αναθεώρηση. Και μετά έχω μια πολύ ειδική ερώτηση. Μου φάνηκε περίεργο, αξιοσημείωτο ότι η κοινή αναθεώρηση αναφέρει μία συγκεκριμένη καταγγελία που έκανα εγώ. Που είχα και στο δικαστήριο. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, ήταν και στι εφημερίδε, είναι δημόσιο. Αλλά είπαν. Αν ας πούμε ήταν τρεις οι καταγγελίες ή οι προσφυγές, θα είχατε βάλει και τα ονόματα και των τριών. Μου τράβηξε την προσοχή αυτό και πολιτικά έχει σημασία που το έχετε βάλει στην έκθεσή σα. Και διερωτώ με γιατί άραγε. Ερώτηση δεύτερη δεν αφορά την κοινή αναθεώρηση, αλλά το νομικό καθεστώς της συμφωνίας με τον Καναδά. Μέχρι σήμερα, τώρα πήρα ένα σημείωμα, δεν έχουμε καταφέρει να διευκρινίσουμε αυτό. Δεν μας έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νομικό καθεστώς της συμφωνίας αυτής και το γεγονός ότι είναι αφήσιμο με κάνει να πιστεύω ότι είναι αρκετά επίγον να προχωρήσουμε σε νέα συμφωνία με τον Καναδά και να εργάζεται η Επιτροπή στο σχέδιο εντολής για την συμφωνία με τον Καναδά. Τρίτον, ζητήσαμε επίσης επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει για ποιο λόγο οι νέοι κανόνες για την ασφάλεια που συνδέονται με τη συλλογή στοιχείων των επιβατών προσωπικών PNR που ζητούν οι ΗΠΑ μία εβδομάδα πριν δημοσιευθεί η κοινή αναθεώρηση. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να μας εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες και πώς θα επηρεάσουν τη χρήση PNR στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτειών. και πότε προτίθεστε να μας τα εξηγήσετε αυτά και να τα διευκρινίσετε. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πότε προτίθεται να μας δώσει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει από τον Νοέμβριο του 2008 σε ψήφισμά μας. Καλά, ε, στο μεταξύ νομικά αυτό πλέον δεν έχει σημασία ε, τυπική γιατί έχουμε περάσει στη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά στην ουσία παραμένουν τα ζητήματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας δώσει εγκαίρως πριν σε νέες διακοπές το πακέτο PNR. Αυτά τα ερωτήματά μου. Ποιοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Oh my God, I frightened you so much, nobody dare. Σας τρόμαξα τόσο πολύ που δεν τολμάει κανείς να πάρει το λόγο και να υποβάλει ερωτήσεις. Brief your remarks, then maybe... Ας ακούσουμε σύντομα τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί έτσι μετά να ε, παρέμβουν και τα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Αλμέιντα. Ε, μετά από όλα αυτά που είπατε, θα χαιρόμουν και εγώ να μην πάρω τελικά το λόγο, αλλά τέλος πάντων. Θα συνοψίσω τις απαντήσεις που είχαμε προετοιμάσει. Για την ε, κοινή ε, έκθεση αναθεώρησης ε, θα έλεγα ότι για την υποστήριξη καταπολέμησης του έγκληματος και της τρομοκρατίας η γέννη ευθυγραμμίζονται με τις υφιστάμενες συμφωνίες. Θεωρούμε ότι τα, υπάρχουν πολύ καλά φίλτρα σχετικά με το Αμερικανικό Nexus και την αποκλειστική πρόσβαση των ΗΠΑ στι 19 κατηγορίες της συμφωνίας, οι κανόνες για την πληροφορία και για την επανόρθωση τηρήθηκαν και... Υπάρχει καλή ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες μόνο όταν συντρέχει ανάγκη και μόνο σε συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις. Θεο, μας ανησυχεί μας ανησυχούν λίγο οι πιθανές ε, λειτουργίες που μπορεί να ε, συγκροτήσουν οι Αμερικανικές ε, αρχές για υπέρβαση του συστήματος και η δυνατότητα δημιουργίας αυτής της ομάδας ad hoc, ad hoc pool, αν μπορώ να το πω έτσι, Θεωρούμε επίσης ότι η διασταύρωση που γίνεται με κάποιες βάσεις δεδομένων θα μπορούσε να συνιστά ένδειξη για πιθανή χρήση και το τονίζω πιθανή χρήση των δεδομένων PNR για λόγους μετανάστευσης και αυτό μας ανησυχεί. Είπα πρέπει να ε, επιφέρουν βελτιώσεις ε, για την αμοιβαιότητα, για την ανταλλαγή πληροφοριών ε, με την ευρωπαϊκή πλευρά ως ανταπόδοση για τις πληροφορίες PNR που παίρνουν για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά αυτή τη χρήση δεν την έχουμε διαπιστώσει μέχρι στιγμή σε μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων, εν γέννη ικανοποιούμεθα από τη μέχρι του εφαρμογή της συμφωνίας από τη ΣΥΠΑ παρότι υπάρχουν κάποιες επικρίσεις που έχουμε συμπεριλάβει στην έκθεσή μας. Για τη συμφωνία με τον Καναδά τώρα, ε, είναι κενή περιεχομένου προς το παρόν, δεν υπάρχει κατάλληλη απόφαση. Και τι γίνεται, το θέμα ε, το χειρίζονται τα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό που λέω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στα κράτη-μέλη να ε, συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις τους ε, ως προς την απόφαση καταλληλότητας adequacy decision ε, για την μεταβίβαση δεδομένων PNR προς τις καναδικές αρχές και γιατί ακόμη δεν έχουμε διαπραγματευτεί μια ουσιαστική συμφωνία με, την, με τον Καναδά. περιμέναμε να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας για να αποφύγουμε τον τρίτο πυλώνα, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπομειστεί πλήρως τα νέα καθήκοντα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε, δεν είμαι και εγώ σίγουρος ε, αν μιλάμε μόνο για PNR ή και για API, αλλά θα έρθουμε σε επαφή με τις Αμερικανικές Αρχές. Η ικανοποιητική απάντηση δεν έχω να σας δώσω, αφού πολύ φοβάμαι προς το παρόν. Για το πακέτο PNR... Τι εννοείται λέγοντας θέρος, ε, ναι, Πάει και μέχρι Σεπτέμβριο, ξέρετε, κατά κάποιους για τον Καναδά, για τις ΗΠΑ ε, ε, και για την Αυστραλία. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε τις εντολές πολύ νωρίτερα από τα Σεπτέμβρη και για την ε, μεταβίβαση διεθνών δεδομένων PNR προς άλλες χώρες του κόσμου το Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Σύστημα PNR θα καθυστερήσει περισσότερο γιατί ε, δύο υπηρεσιακά μας ενημέρωσαν ότι χρειάζεται νέα αξιολόγηση αντικτύπου για να στοιχειοθετηθεί η πρόταση, θα διγοτομηθεί η πρόταση. Θα έχουμε τις τρεις εντολές και την ανακοίνωση ελπίζουμε το Σεπτέμβριο... αλλά το σύστημα PNR λίγο αργότερα, στα τέλη του τρέχοντος, στις αρχές του επομένου. Ωραία. Για να συνοψίσω, ε, summer break, λέει mid-July, άρα μέσα Ιουλίου. Το λέει σαφώς μέσα στην ανακοίνωση. Και ελπίζω να έχουμε σύντομα τις απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι οι κανόνες ασφαλείας ε, των ΗΠΑ μιλάνε για ε, data mining, ε, που, κανόνες που άρχισαν να ισχύουν το Φεβρουάριο και σε λίγο αύριο είναι Ιούνιος. Δεν μπορείτε να κινηθείτε ταχύτερα. Περιμένουμε γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εμάς και προς το Συμβούλιο για τα ε, ζητήματα που αναφέραμε στο ψήφισμα του Νοεμβρίου του 2008 και για τα οποία δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση. Ο κύριος Άλμπερ. Θα προσπαθήσω να είμαι και πάλι σύντομος. Υπάρχει ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Το εξής. Εμείς πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε πιο πέρα στο πακέτο PNR, γιατί μπορεί να μην έχουμε αναγνωρίσει ακόμα το πρόβλημα, αλλά το έχει τονίσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο. Για μας, οι συμφωνίες που προτείνονται, όπως τις έχουμε στα χέρια μας, είναι απαράδεκτες. Αυτό προσπαθώ να σας πω εδώ και το έχω διαπιστώσει και κατά πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή χρειαζόμαστε νέες διαπραγματεύσεις. Αλλά ως Κοινοβούλιο δώσαμε την ευκαιρία οι κείμενες συμφωνίες να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, παρόλο που πολλοί από εμά εδώ μέσα θεωρούμε ε, ασύμβατες με τις συνθήκες τις συμφωνίες αυτές. Δηλαδή θα πρέπει κάθε φορά να εξηγούμε στους πολίτες γιατί αφήνουμε να ισχύουν συμφωνίες χωρίς να τις πάσουμε ε, συμφωνίες με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένες. Και επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι αυτό είναι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να έχει τη δυνατότητα το Κοινοβούλιο να ξέρει και γρήγορα ε, ποια θα είναι η νέα συμφωνία και να ασχολείται με τη νέα συμφωνία και όχι να παραμένουμε ε, σε αυτό το προσωρινό και να μην έχουμε και την αίσθηση ότι χρονοτριβούμε και το αναβάλουμε και κολλησιεργούμε και καλό Οκτώβρη και καλό Νοέμβρη θα ερχόμαστε να τα συζητάμε στο Κοινοβούλιο και να συνεχίζει να εφαρμόζεται. Από πότε είναι αυτό? Από την 1η Πρώτου 2007 κιόλα. Χωρίς να συμφωνεί και χωρίς να έχει ψηφίσει έστω και ένα κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα είναι αφόρητες καταστάσεις αυτές. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Επιτροπή Εσωτερικών και Ελευθεριών, όπως τη λέμε, να έχουμε ε, γνωμοδότηση, να έχουμε απόφαση του Δικαστηρίου ε, για το τι συμβαίνει με αυτές τις συμφωνίες που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Δεν θεωρώ σωστές αυτές τις χρονοτριβές. Χρειάζεται να κινηθούμε πολιτικά. Ευχαριστώ, κύριε Φως. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω, όπως είπατε, αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Οι δύο, συμφωνώ και με τους δύο και ιδιαίτερα με τον Γιάνν Φίλιπ Άλμπρεχτ που μίλησε τελευταίος. Θα ήθελα να σας πω ότι για τον Καναδά δεν με ικανοποιεί καθόλου αυτό που συμβαίνει. Αν κατάλαβα σωστά ότι τώρα λέει θα κατακαιρματιστούμε, θα χωριστούμε θα κράτη-μέλη. Μα δεν είχαμε αυτή την πρόθεση αρχικά. Και δεν είναι καθόλου σωστό αυτό. Θα πρέπει το συντομότερο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. αναβάλαμε τη συμφωνία με την Αυστραλία και με τη ΣΥΠΑ και ε, ε, νομίζω ότι φταίμε το, εμείς γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Κοινοβούλιο, δεν ξέρω ποιος, ε, θα πρέπει γρήγορα να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα έγγραφα αυτά, έτσι ώστε και στη διατλαντική σχέση μας ή τη σχέση μας με την Αυστραλία να είμαστε σωστοί. Και ένα τελευταίο Μήπως θα μπορούσαμε να πιέσουμε να μην έχουμε διπλή συλλογή στοιχείων. Θα ήταν και αυτό καλή κίνηση και πρόοδος. Ευχαριστώ. Κυρία Ernst. Ναι, και εγώ πολύ σύντομα. Εκπλήσωμαι από αυτά που ακούω για τον Καναδά συνολικά. Είναι αξιοσημείωτα σε ποια κατάσταση έχουμε περιέλθει. Και εγώ θεωρώ λάθος να τα χωρίσουμε στα κράτη-μέλη αυτά. Εμείς ζητούμε νέες διαπραγματεύσεις και θέλω να θυμίσω κάτι που είχαμε δεχτεί τον Απρίλιο, ένα ψήφισμα που ζητάει και ελάχιστε προδιαγραφές, ξεκάθαρα, που θα πρέπει να επεξεργαστούμε μία προς μία. Και προς το παρόν τα βλέπω όλα πάρα πολύ θολά και συγκεχημένα και ασαφή. Πίεση πρέπει να ασκήσουμε. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ κύριε Ζήπελ. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν, αλλά θεωρώ σημαντικό να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τις ε, ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Και πού δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε πει επανειλημμένα, δεν θέλουμε τρεις-τέσσερις συμφωνίες που να διαφέρουν πάρα πολύ στις λεπτομέρειες τους, αλλά θέλουμε να έχουμε μία συμφωνία προς όλους. Και για μένα το καλοκαίρι δεν τελειώνει το Σεπτέμβριο. Τι είναι αυτά τώρα τα χρονοδιαγράμματα και τα ημερολόγια. Στο δικό μου ημερολόγιο το αργότερο Αύγουστο τελειώνει το καλοκαίρι. Αφήστε δε που θεωρώ ότι πρέπει πριν τις ελληνές διακοπές να έχουμε ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Μα ξέρετε δεν είναι και καινούργια αυτά τα πράγματα με τα PNR. Τι κάνουμε, παίζουμε τις καθυστερήσεις εδώ τώρα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θέλουμε και ε, πώς θα λάβουμε υπόψη μας στο κοινοβούλιο. και κατά πόσο αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή του σοβαρού εγκλήματος. Καθόλου δεν είναι σαφές αυτό. Και θα πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα από την Επιτροπή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μας ικανοποιεί η κατάσταση αυτή. Να χρησιμοποιούνται για τελευ... τε... τελείως άσχετους ε, σκοπούς μέχρι την αρχή, όχι το τέλος των θερινών διακοπών θέλουμε να έχουμε τη νέα πρόταση για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε. με πάσα σοβαρότητα δηλώσαμε την πρόθεσή μας να εκπονήσουμε αυτές τις τρεις εντολές και την ανακοίνωση. Μπορεί να καθυστερήσουμε λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο. Ορισμένε φορές ε, ε, δεν κατορθώνουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Θα τις πάρετε τις τρεις εντολές και την ανακοίνωση το ταχύτερο δυνατόν. Ευελπιστούμε μέσα στο καλοκαίρι. Ή το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη το αργότερο. Ε, τι να σε εξηγήσω τη διαδικασία, τα γραφειοκρατικά στάδια που χρειάζονται για την απόκτηση των εντολών έχουν συνταχθεί οι εντολές, έχουν φύγει από την υπηρεσία μου και ανεβοκατεβαίνουν, πηγαίνουν αριστερά δεξιά σε όλες τις υπηρεσίες, θα σας φτάσουν και σας, ε, είμαστε πάρα πολύ σοβαροί, έχουμε την πρόθεση να σας υποβάλουμε προς τον κύριο Άλμπρεχτ θα πω ότι ελπίζουμε να είμαστε πιο γρήγοροι από το δικαστήριο. Ε, ε, δηλαδή πιο γρήγορα θα πάρετε τις εντολές παρά την ε, απόφαση του δικαστηρίου. Τώρα, δεν υπάρχει διαχωρισμός. Η ανακοίνωση και οι τρεις εντολές θα παραμείνουν μαζί στο ίδιο πακέτο. Σας μίλησα για διχοτόμηση σε σχέση με το, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε την ανακοίνωση νωρίτερα, ότως ώστε να μην βρεθείτε πρώτα τελεσμένο και να δεχτείτε κάτι που πήρατε τελευταία στιγμή. Δηλαδή θα σας δώσουμε την ευκαιρία να επηρεάσετε τις εξελίξεις. Με τον Καναδά ε, δεν είχαμε εντολή πέρσι δεν γινόταν ε, ε, γιατί ακόμη δεν είχε τι νέε εξουσίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει τη συνθήκη Λισαβόνα και αυτό είναι ο μόνο λόγο που δεν κάναμε τίποτα πέρυσι με τον Καναδά. Πρόεδρος, ε, να κάνω κάποιες καταλεκτικές παρατηρήσεις με την ιδιότητα της εισηγήτριας. Ε, παρακαλούμε, εργαστείτε ταχύτατα. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Και όπως σωστά σας υπενθύμησαν ε, οι συναδελφοί σας, έχουμε δώσει πολύ χρόνο. Μπορούμε, ξέρετε, να ψηφίσουμε. Έχουμε και άλλη εναλλακτική. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ναι, επαχθεί γραφειοκρατικέ διαδικασίε, αλλά μην προτάσετε αυτό το επιχείρημα σε τόσο καθυστερημένο στάδιο. Για το SWIFT σε 10 μέρε τα καταφέρατε. Ε, και με λιγότερα μέλη τώρα η νέα επιτροπή νομίζω μπορεί να ε, ε τα καταφέρει γρηγορότερα. Και αν βιαστείτε με τόσε πολλέ αποφάσει για να προλάβετε πριν την 1η Δεκεμβρίου, γιατί λοιπόν για τον Καναδά ούτε καν μα ενημερώσατε, δηλαδή η μεταφορά καταστάσεων επιβατών αυτή τη στιγμή προ τον Καναδά δεν έχει ε, κρατεά νομική βάση. Αυτή είναι η κατάσταση. Εσεί εγνέφετε αρνητικά. Εγώ είμαι πεπισμένη όμω ότι έχω δίκιο. Δεν θέλω να σα δυσκολέψω, αλλά πρέπει επιγόντω να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να γίνει αυτό πριν τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Αυτή την ημερομηνία ε, είχαμε ζητήσει, αυτή θα στοχεύσουμε λοιπόν. Δεύτερον, όλες οι ερωτήσεις που ακούσατε στη συζήτηση και όλες οι γραπτές ερωτήσεις ε, που πήγαν στην υπηρεσία σας ε, περιμένουν απάντηση, γραπτή απάντηση από την υπηρεσία σας και η αναφορά στο όνομά μου είναι ένα από αυτά τα θέματα για τα οποία περιμένω απάντηση. Νομίζω κλείσαμε τώρα το θέμα PNR και την μερίσια διάταξη για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε στις 9, έτσι. Είναι μεικτή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γυναικών. Αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστώ.